<clears throat> Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην 10η Σύνοδο της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Σερβίας. Έχουμε διερμηνία στα αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά και σερβικά. Τα σερβικά τα έχετε στο κανάλι 25. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε κροατικά. <laughs> Δεν ξέρω γιατί. Έχουμε πάντως, ε, για κάποιο λόγο, τη λεγόμενη παθητική διερμηνία. Από τα κροατικά στις άλλες γλώσσες. Καλωσορίζω ειλικρινώς τα μέλη και των δύο αντιπροσωπιών και όλος ιδιαίτερος τους φίλους από τη Σερβία διότι πήραν μια πτήση πάρα πολύ νωρί σήμερα από το Βελιγράδι, αλλά τους βλέπω φρέσκους φρέσκους. Φαντάζομαι ότι θα εργαστούμε ως συνήθως. Να καλωσορίσω επίσης τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, τον Ιουκοσλαβ Μιλατσέτς, σύμβουλο του Υπουργού Ευρωπαϊκής πολιτικής εκ μέρους της κυβέρνησης της Σερβίας. Να καλωσορίσω επίσης τον κύριο Τσάμπα, Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Αποτελεί αυτό καινοτομία στην Επιτροπή μας, αλλά η παρουσία αυτή είναι ευπρόσδεκτη στις εργασίες μας. Επίσης, τον κύριο Χρήστο Μακρίδη, επικεφαλής της μονάδας της Digineer για την Σερβία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως και τέλος, τον κύριο Ράμπολτ, από τη Διεύθυνση Δυτικών Βαλκανίων, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σας ενημερώνω επίσης ότι Έχουμε εδώ εκπαιδευόμενους που θα μας παρακολουθούν. Τους ε, καλωσορίζω ειλικρινώς. Διότι τα νέα αυτά παιδιά είναι το μέλλον μας και πρέπει να τους φροντίσουμε. Πριν ε, έλθουμε στην ημερήσια διάταξη, στα θέματα ουσίας, ε, κάποια τυπικά έγκριση ημερήσια διάταξη. Σχόλια για την ημερήσια διάταξη, για το σχέδιο μάλλον ημερήσια διάταξης. Όχι, από ό,τι βλέπω. Οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Δεύτερον, έγκριση σχεδίου πρακτικών της ένατης συνεδρίασής μας, που έγινε στις 29 και 30 Οκτωβρίου στο Βελιγράδι το 2018. Η Γραμματεία έχει διανύμει σχέδια πρακτικών με ενημερώνουν ότι δεν έχει ζητήσει κάποιος τροποποίηση εντός της προθεσμίας. Οπότε, θέλει κανείς να μιλήσει για τα δύο αυτά θέματα. Όχι. Οπότε, εγκρίνουμε και την μεσή διάταξη και τα πρακτικά. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, επιτρέψτε μου να διατυπώσω ορισμένε παρατηρήσεις ε, θα χαριστώ λίγο περισσότερο χρόνο. Είναι η τελευταία μας συνεδρίαση. Ε, δεν θέλω να προκαλέσω νοσταλγία σε κανέναν, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργώς την πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τάσεται υπέρ της ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να εξασφαλίσει η ανάπτυξη και ευημερία. Θεωρώ τι εργασίε μα, τι εργασίε τη Επιτροπή μα, σημαντική συμβολή στη διαδικασία αυτή. Όπω γνωρίζετε, πρόκειται για την τελευταία συνεδρίασή μα στα πλαίσια τη παρούση θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014-2019. Προσεχώ έχουμε εκλογέ τέλη Μαΐου προσεχώς. Οπότε είναι και η τελευταία φορά που συναντάτε τη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρουσία της σύνθεση και σίγουρα είναι και τελευταία φορά για μένα που συμπροεδρεύω την Διακοινοβουλευτική Επιτροπή διότι δεν είμαι υποψήφιος, δεν θα είμαι υποψήφιος στις προχείς εκλογές. Ελπίζω εν τούτης, ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργώ την πολιτική διεύρυνση και να υποστηρίζει βεβαίω και την ένταξη τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω έπραξε άλλωστε και το παρόν Κοινοβούλιο. Όπω γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την έκθεση τη Κομισιόν για τη Σερβία στην Ολομέλεια του Νευρίου, όπου παραλαμβάνουμε τη θέση μα επί των διαπραγματεύσεων ένταξη και διατυπώσαμε και συστάσεις για τα βήματα που είναι απαραίτητα για να αντιμετωπιστούν οι μείζονες προκλήσεις και να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί και την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την πρόοδο που επιτέλεσε η Σερβία σήμερα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Σερβία προχωρά οικονοποιητικά στις διαπραγματεύσεις εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την προσήλωση της Σερβίας στον δρόμο της ένταξης και συγχαίρουμε τη Σερβία για τις προσπάθειες της να υποστηρίξει την στρατηγική αυτή απόφαση και στην σερβική κοινή γνώμη. 55% των Σέρβων, σύμφωνα με πρόσφατε δημοσκοπήσει, υποστηρίζουν την ένταξη τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τούτη όμω, σύμφωνα με τι ίδιε δημοσκοπήσει, 67% των Σέρβων δεν έχουν ακούσει ποτέ το παραμικρό για κάποιο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα. Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος, ο σημαντικότερος δωρητής στη Σερβία. 7 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν με τη μορφή επιχορηγήσεων ιδανείων τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτή είναι η επένδυσή μας στο μέλλον της Σερβίας. Οι Σέρβοι δικαιούνται να γνωρίζουν λοιπόν. Συνεπώς σας ενθαρρύνουμε θερμά να ενημερώσετε τους Σέρβους πολίτες για τα έργα αυτά. Γιατί μπορεί να μιλάμε για την διεύρυνση, αλλά χρειάζεται να είμαστε και σαφείς περί των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που έχει πορεία αυτή. Εκφράζω επίσης την ικανοποίησή μου για την πρόοδο που σημείωσε η Σέρβια στην ανάπτυξη μιας λειτουργικής ελεύθερης οικονομίας, για περισσότερη ανάπτυξη, η περισσότερη μακροοικονομική και νομισματική σταθερότητα. Η προσπάθεια αυτή έχει ως απότοκο τη μείωση της, τη μείωση της ανεργίας. Επίσης, είμαστε υπέρ της δημοσιονομικής εξυγίανσης, αποφασιστικής σημασίας για να αποκτήσει ο κόσμος εμπιστοσύνη στην οικονομία. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο προπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης από έλλειμμα 6,6% που παρουσίαζε σε σχέση με το ΑΕΠ, πέτυχε πλεόνασμα 1,2%. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για την πολιτική χωρίς αποκλεισμούς που υιοθετείται στον τομέα των μέσων. Καλή βεβαίω η πολιτική, είναι πολιτική μας που πρέπει να υλοποιηθεί στην πράξη. Στείλαμε επίσης το μήνυμα συναφώς ότι η βία και ο εκφοβισμός κατά δημοσιογράφων δεν έχουν χώρο σε μια χώρα η οποία επιθυμεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι Πρόβλημα το οποίο δυστυχώ οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, μέλη ήδη δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν κάποια πρώτα βήματα με τη μορφή τη σύλληψη των υπευθύνων ορισμένων κρουσμάτων Βία, όπω γνωρίζετε όμω η Επιτροπή για το συμπέρασμα ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδο για τέταρτη συνεχή χρονιά στον τομέα τη ελευθερία τη έκφραση. Μάλιστα η Σερβία έπεσε 10 θέσει την Παγκόσμια Κατάταξη Ελευθερίας του Τύπου του 2018 σε σχέση με το 2017. Αυτή η έλλειψη πρόοδου αποτελεί πηγή ανησυχίας, όπως καταλαβαίνετε για μας. Η Σερβία είναι μια πλουραλιστική χώρα όσον αφορά τα μέσα. Παρέχει αρκετές διασφαλίσεις στην προστασία των δημοσιογράφων συμπεριλαμβανομένων των τοπικών μέσων. Εάν χρειάζεται βοήθεια στην ενημέρωση όσον αφορά τη γενικότερη αντιμετώπιση των δημοσιογράφων και των μέσων, ε, Ευχαριστώ να σας βοηθήσουμε. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είναι όλο και πιο σημαντικό λόγω των πρόσφατων διαδηλώσεων τους τελευταίους τέσσερις μήνες στη Σερβία και την πρόσφατη βίαιη εισβολή στην κρατική ραδιοφωνία τηλεόραση. Τα γεγονότα αυτά δηλώνουν για άλλη μια φορά ότι χρειάζεται ευρύτερος διάλογος κατά της βίας. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίε με το περιεχόμενο των ειδήσεων, αλλά αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με βία και εκφοβισμό των δημοσιογράφων. Ορθώ δήλωσε ο πρεσβευτή σα, κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία την περασμένη εβδομάδα στι Βρυξέλλε, ότι η ακυρότητα των μέσων είναι ιερή, αλλά να προσθέσω και εγώ από την πλευρά μου ότι ακόμα πιο ιερή είναι η ελευθερία των μέσων και η ανεξαρτησία της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Όσον αφορά τις ε, τρέχουσες διαδηλώσεις, να τονίσω ότι όλα αυτά είναι μέρος μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Είναι συνήθις της δημοκρατίας μας. Είναι δικαίωμα των πολιτών να κινητοποιούνται ειρηνικά. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να αποφεύγουν από πράξεις βίας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η κυβέρνηση της Σερβίας να κάνει κάτι για να καθισχάσει τις ανησυχίες των πολιτών της. Εμείς ως κοινοβουλευτικοί παρακολουθούμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Βουλή της Σερβίας στο νομοθετικό και ελεγκτικό της έργο, κάτι το οποίο οδήγησε ορισμένους βουλευτές να μποϊκοτάρουν τη λειτουργία της Βουλής. Αυτό που μας ενισχύει είναι το υπερβολικό πλήθος κατεπηγουσών διαδικασιών αλλά και άλλες πρακτικές που δεν ε, βοηθούν βεβαίως, ε, δεν είναι υπέρ της ποιότητας του νομοθετικού έργου. Το Κοινοβούλιο είναι κέντρο δημοκρατικού διαλόγου. Εκεί τόσο η συμπολίτευση όσο και η αντιπολίτευση προσπαθούν να εξεύρουν από κοινού λύσεις και απαντήσεις για αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Ενθαρρύνω όσο πιο θερμά μπορώ την κυβέρνηση να εξασφαλίσουν συνθήκες ικανοποιητικού διαλόγου. Γνωρίζω ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της ΑΦΕΤ ε, τέλη Φεβρουαρίου υπό τον ε, κύριο Μακάλιστερ στη Σερβία έγινε μια σχετική συζήτηση και έγινε αναφορά στη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διευκολύνει την επικοινωνία των κομμάτων για να καταλήξουν από κοινού σε κάποιο κώδικα δεντολογίας και κανονισμό για τη Βουλή. Ε, πρόκειται για υποστήριξη την οποία μπορεί να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των λεγόμενων διαλόγων Ζαν Μονέ. Ήδη έχει αξιοποιηθεί αυτό ο διάλογο, ε, όπω για παράδειγμα στην Βόρεια Μακεδονία και στην Ουκρανία. Οπότε παρακαλώ εξετάστε και αυτό το ενδεχόμενο να βοηθήσουμε τους φίλους μας στη Σερβία όσον αφορά τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Με βέβαιο ότι ήδη γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και αποκλείεται να εισαγάγει διμερείς διαφορές στο εσωτερικό της. Εμείς θέλουμε και οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να προσπαθούν να βρουν μια αμοιβαίως δεσμευτική νομική συμφωνία. Αυτό θα είναι πρώτα απ' όλα προς το συμφέρον όλων των πολιτών της περιοχής. Το Βελιγράδι και η Πρίστινα οφείλουν να καταλήξουν σε συμφωνία με την οποία θα επιλύσουν όλα τα εκρεμή ζητήματα πριν γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να καταστεί αυτό δυνατόν και η Πριστινά και το Βελιγράδι πρέπει να δημιουργήσουν το κλίμα το οποίο θα καταστεί το διάλογο δυνατό. Και το πρώτο βήμα προκειμένου είναι οι αρχές της Πρίστινας να καταργήσουν τους δασμούς 100% ε, επί εμπορευμάτων που παράγονται στην Σερβία. Όσον αφορά την ιδέα που ακούμε να συζητείτε όσον αφορά τη διόρθωση των συνόρων και την ανταλλαγή εδαφών, επαναλαμβάνω την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο οφείλουν να παραμείνουν πολυεθνικέ χώρε και θα μπορούσαμε να δεχθούμε οποιαδήποτε συμφωνία με την προπόθεση ότι την χάνει κοινή αποδοχή και ότι συμβαδίζει, συνάδει με το διεθνέ δίκαιο και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη γενικότερη σταθερότητα στην περιοχή. Τέλο, να και τα κλείδι ότι επιθυμούμε να δούμε περισσότερη πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις, τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην Σερβία, ιδιαίτερα στον τομέα του κράτους δικαίου, κάτι το οποίο αποτελεί και προϋπόθεση για το άνοιγμα νέων κεφαλαίων. Στην έκθεση της Freedom House του 2018, η Σερβία ήταν η μόνη χώρα η οποία χαρακτηριζόταν ως ελεύθερη, συνολικά χωρίς ε, επιφυλάξει. ενώ οι άλλε πέντε χώρε των Ιντερικών Βαλκανίων χαρακτηρίζονταν ω μερικώ ελεύθερε. Και όμω το 2019, στην, έκθεση, στην έκδοση μάλλον τη ίδια έκθεση, η Σερβία έπεσε από το ελεύθερη σε μερικώ ελεύθερη. Και μάλιστα είναι τέταρτη πλέον στον καταλόγο των χωρών ε, που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση το 2000, σε σχέση μάλλον με το 2018. Ε, πρόκειται για επαναχώρηση στον τομέα αυτό και το λέω αυτό διότι μπορεί να έχει απογοητευτεί η Σερβία όσον αφορά την, βραχία, την αργή πρόοδο στο άνοιγμα κεφαλαίων, αλλά αυτό είναι φυσικό. Όσο οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου δεν προχωρούν επαρκώς, όσο και η πρόοδος στην εξομαλύση των σχέσεων με την Πρίστινα. Χωρί σαφή πρόοδο στα κεφάλαια 23 και 24, το πράγμα δεν προχωράει. Και αυτό είναι ένα σαφέ μήνυμα τόσο για τη Σερβία, όσο και για τι άλλε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτή ήταν η σύντομη εισαγωγή μου, κυρίες και κύριοι. Και κλείνω όπως είπα με απόλυτη ειλικρίνεια ότι πραγματικά ήταν για μένα χαρά και τιμή να συμπροεδρεύω τα τελευταία δέκα χρόνια. Ήταν μεγάλη μου χαρά που συνεργάστηκα με όλους σας. Έκανα φίλους εδώ. Φίλες που θα κρατήσω και στο μέλλον με τους Σέρβους συνδέλφους. Οπότε δίνω τον λόγο στο σημείο αυτό, στον κύριο Όρλιτς τον συμπρόεδρο. Για τις δικές του εισαγωγικές παρατηρήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης, ε, αγαπητοί εκπρόσωποι τη Σερβικής Κυβέρνησης, μέλη του Σερβικού Κοινοβουλίου και από τους υπόλοιπους ε, συμμετέχοντε στη συνεδρίαση. Επιτρέψτε μου να σα πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σε αυτή τη συνεδρίαση και που έχουμε γενικά αυτή τη συνεδρίαση. Είναι η δέκατη και θα συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο κύριος Κούκαν. Αυτή η δέκατη συνάντηση λοιπόν λαμβάνει χώρα ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι είναι η τελευταία συνάντηση κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής ε, θητείας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική για όλους μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να στραφώ στους ε, αγαπητούς συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προς εσάς κύριε Κούκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, για τη στήριξη, καθ' τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Η συνεργασία μαζί σας ήταν για μας ένα προνόμιο και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Το γνωρίζετε, αλλά θα ήθελα να επενθυμίσω ότι η φιλία αυτή ξεπερνά τα όρια της δουλειάς που κάνουμε εδώ και πάντα στο πρόσωπό μας θα βρίσκεται πραγματικούς φίλους. Από την πρώτη συνάντηση του 2013 μέχρι και σήμερα, που είναι η δέκατη συνάντηση, αυτό ισχύει. Όλα όσα καταφέραμε να πετύχουμε μέχρι τώρα οφείλονται μέρη και στη δική σας ε, προσπάθεια και συμβολή. Σίγουρα και εμείς ε, θα βρούμε συμμάχους ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλες οι μελλοντικέ μας συναντήσεις θα αποτελέσουν ένα βήμα προς το μέλλον, προς την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας για το 2025. Γνωρίζετε ότι η στήριξη για την ένταξη τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερή, είπατε και εσεί ότι είναι 55% στη Σερβία. Αυτό προκύπτει από το Ευρωβαρόμετρο. Μπορείτε να το βρείτε ε, στο Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σερβίας και στον σχετικό ιστότοπο. πρέπει πρώτα να δούμε τι ακριβώς χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να προβάλλουμε το έργο της. Βάσει της ίδιας δημοσκόπησης μπορώ να σας πω ότι οι Σέρβοι πολίτες σήμερα για πρώτη φορά μιλούν για τις ε, ευρωπαϊκές χώρες και τις ευρωπαϊκές χορηγίες και δωρεές. Κατανοούν λοιπόν πλέον οι Σέρβοι πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά σημαντικός ε, σύμμαχος, ότι οι Ευρωπαίοι είναι φίλοι τους. Φυσικά και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία, είναι κοινό μας ε, καθήκον και για μας τους δημόσιους λειτουργούς στη Σερβία, αλλά και οι Ευρωπαίοι φίλοι μας που εξηγούν στους πολίτες μας και έτσι αυξάνουν την στήριξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Σερβίας. Γιατί αποστέλουν το σωστό μήνυμα την κατάλληλη χρονική στιγμή. Η τάση από το 2016 και μετά υφίσταται και συνεχίζει να υπάρχει. Είναι μια θετική λοιπόν δυναμική. Είναι σημαντικό ε, που η Ευρωπαϊκή, μάλλον σημαντικό Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να υποστηρίζει τα Δυτικά Βαλκάνια, όπως είδαμε το 2018. Η ένταξή μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο υπαριθμόν ένα στόχος μας καταβάλουμε προσπάθειες ε, για την επίτευξη των στόχων μας ε, όπως ε, προβλέπονται στο πρόγραμμα δράσης προκειμένου να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο που είναι η ένταξή μας το 2025. Βλέπετε λοιπόν ότι η Σερβία αυτή τη στιγμή διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική. Δεν το λέμε εμείς αυτό οι Ευρωπαίοι φίλοι μας το λένε. Και μία σόφρονα πολιτική την οποία ακολουθούμε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και μεγαλύτερη από τις προκλήσεις είναι αυτή του κοσυφοπεδίου. Προβλέπετε, βέβαια και ειδικό σημείο στη Μέση διάταξη για αυτό το ζήτημα. Θα σταθώ λοιπόν στη συνέχεια και σε όλα τα σημεία που θίξατε εσείς κύριε Κούκαν στα εισαγωγικά σας σχόλια. Θα ήθελα όμως να πω ότι η σημερινή συνάντηση θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα πλουραλισμού, όπως είπατε κι εσείς. Θα πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, να μιλήσουμε για τα σχέδιά μας, τις προσδοκίες μας, να συμφωνήσουμε επί ορισμένων σημείων και βέβαια να παρουσιάσουμε τα επιχείρηματά μας και για τα σημεία στα οποία διαφωνούμε. Η κριτική πάντα είναι καλοδεχούμενη στις συναντήσεις μας έτσι κι αλλιώς. Η κριτική βέβαια εύκολα μπορεί να αποφευθεί όταν δεν κάνει κανεί τίποτα, αλλά εμεί ξέρετε ότι δεν ακολουθούμε αυτή την άγουσα, Αντιθέτω, θέλουμε να έχουμε έναν πολύ ποιοτικό διάλογο. Και χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί σε πολλά συμφωνούμε. απόδειξη είναι το κείμενο που έχετε λάβει, που έχουν αποστέλει δύο συμπρόεδροι. Αν το διατρέξετε, ελπίζω να μείνετε ικανοποιημένοι από τη διατύπωση στην οποία καταλήξαμε σε επίπεδο Προεδρείου πριν από αυτή την συνεδρίαση. Και ελπίζω να συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή προκειμένου να ενταχθεί η Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συμπρόεδρε. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3 τη εμείς διάταξη που αφορά την κατάσταση ως προς τις διαπραγμα... διαπραγματεύσει ε, τη Σερβίας παρουσία εκπροσώπων ε, της Σερβικής Κυβέρνησης, ε, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιούγκοσλαβ Μίλατσιτς, ε, σύμβουλο του Υπουργού Ευρωπαϊκής Ένταξης, για να μας παρουσιάσει την οπτική γωνία της Σερβικής Κυβέρνησης. Ευχαριστώ, κύριε Κούκαν κύριε Όρλιτς. Εκπρόσωποι της ε, Προεδρίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, Σερβικής ε, Βουλής. Θα ήθελα να σας δώσω μια σύντομη εικόνα της κατάστασης ό,τι αφορά τις πρωτεξιακές διαπραγματεύσεις. Θα είμαι σύντομος αλλά θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω και τα πολιτικά κριτήρια που άπτονται του κράτους δικαίου ε, και της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Πελεγραδίου και Πρίστινας. Όπως γνωρίζετε, η Σερβική Δημοκρατία έχει ανοίξει 16 κεφάλαια και προσωρινά έχουν κλείσει δύο από αυτά. Το 25 έρευνα και επιστήμη και το 26 ε, παιδεία και πολιτισμό Θα τέλη του 2016 και αρχέ του 17. Τα αναπομείναντα είναι ε, αυτό των δημοσίων συμβάσεων που άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 2016, το 6 του εταιρικού δικαίου τον Δεκέμβριο του 2017, κεφάλαιο 7 ε, πνευματικά δικαιώματα τον Ιούνιο του 2017, το κεφάλαιο 13 αλληλεία τον Ιούνιο του 2018, το 17 οικονομική και νομισματική πολιτική και 18 στατιστικά στοιχεία τον Δεκέμβριο του 2018. Το 20 επιχειρηματικότητα και επιχειρηματική πολιτική. 23 και 24 κράτος δικαίου τον Ιούλιο του 2016. Το κεφάλαιο 29 Τελωνιακή Ένωση τον Ιούνιο του 2017. Το 30 οικονομικές σχέσεις ε, με τρίτες χώρες. 32 και 33 δημοσιονομικές ε, διατάξεις και εποπτεία και άλλα ζητήματα το Δεκέμβριο του 2015. Πέραν τούτων, η Σερβική Δημοκρατία έχει προετοιμάσει ενεργά διάφορα σημεία διαπραγμάτευσης. Πέντε από αυτά έχουν υποβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Προεδρία και άπτονται των εξή κεφαλαίων. Κεφάλαιο 2. Ελευθερία κυκλοφορία των ε, εργαζομένων. Είναι κάτι το οποίο υιοθετήθηκε ως ε, θέση διαπραγμάτευση τον Ιούλιο του 2018 και επίσημα επευλήθη προς την Επιτροπή στις 20 Ιουλίου του περασμένου έτους. Κεφάλαιο 4. Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. μια θέση πραγμάτευσης που υιοθετήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2018 και επιβλήθη πάλι το Σεπτέμβριο του 2018. Κεφάλαιο 9, δημοσιονομικές υπηρεσίες, χρήματα οικονομικές υπηρεσίες, 14, πολιτική μεταφορών και 21, διευρωπαϊκά δίκτυα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν υποβληθεί προς την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και περιμένουμε θετικές απαντήσεις για το άνοιγμα νέων ε, κεφαλαίων για το στάδιο των τεχνικών διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο του τρέχοντος. Και άλλα κεφάλαια είναι έτοιμα και βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασιών, όπου το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει τις εκθέσεις από την εξέταση και μετά η Σερβική Δημοκρατία πρέπει να υποβάλει θέσει διαπραγμάτευση. Έχουμε δύο τέτοια κεφάλαια, το 10, ε, μέσα ενημέρωση ε, και κοινωνία τη πληροφόρηση και 28, προστασία καταναλωτών και υγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλέσει τη Σερβική Δημοκρατία να υποβάλει τις ε, θέσεις της για το κεφάλαιο 10 στις 20 Ιουλίου. Υπευλήθη λοιπόν ένα προσχέδιο τον περασμένο Ιούλιο. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 28, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει παρατηρήσεις επί της θέσης που υπευλήθη τον Νοέμβριο του 2017 και το τελευταίο προσχέδιο κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2018. Και σε αυτή τη βάση λάβαμε παρατηρήσεις στις 14 Μαρτίου του 19. Τα κεφάλαια για τα οποία η Επιτροπή έχει υποβάλει τα αποτελέσματα εξέτασης είναι το 27, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, και εμείς στείλαμε το πρώτο προσχέδιο της διαπραγματευτικής μας θέσης τον Ιούνιο του 2018. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε τις παρατηρήσεις της στις 30 Ιουλίου του 2018. Στη συνέχεια υποβάλαμε και δεύτερο προσχέδιο διαπραγματευτικής θέσης το Δεκέμβριο του 2018. αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να οριστικοποιήσουμε αυτή την πλατφόρμα διαπραγμάτευσης. Στις περισσότερες ε, περιπτώσεις ελάβαμε benchmarks για μια σειρά κεφαλαίων, εννέα τον αριθμό. Το κεφάλαιο 1, ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, όπου έχουμε δύο κριτήρια αναφοράς για το άνοιγμα του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο 3, ελευθερία εγκατάστασης και παροχή υπηρεσιών, όπου έχουμε ένα κριτήριο αναφοράς. Το κεφάλαιο 8, πολιτική ανταγωνισμού, όπου έχουμε 6 κριτήρια αναφοράς για το άνοιγμα. Κεφάλαιο 11, γεωργία ε, και αγροτική ανάπτυξη, 2 benchmarks εδώ. Κεφάλαιο 12, ασφάλεια τροφίμων και φυτογενομική πολιτική, δύο κριτήρια αναφοράς. Κεφαλαίο 15, ενέργεια, με δύο σημεία αναφορά. Το κεφάλαιο 16, φορολογία, με ένα σημείο αναφορά, Κεφάλαιο 19, κοινωνική πολιτική και απασχόληση, ένα κριτήριο αναφοράς. Και κεφάλαιο 22, περιφερειακή πολιτική και συντονισμός ε, διαδοτικών ε, μέσων, όπου και πάλι έχουμε ένα κριτήριο αναφοράς για το άνοιγμα. Επιπλέον έχουμε δύο κεφάλαια για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε εκθέσεις μετά τη διαδικασία εξέτασης, αλλά ακόμα περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα, την τελική έκθεση, για το 31 εξωτερική ασφάλεια και 34 θεσμικά όργανα. Έτσι έχετε μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης. Τα γνωρίζετε φαντάζομαι αυτά, αλλά εφόσον έχουμε εκπροσώπους ε, από διάφορους τομείς ενδιαφέροντος, ήθελα να τα παρουσιάσω συνολικά. Τώρα, να πω και δύο λόγια για τα πολιτικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με την εξομάλυση των σχέσεων με την Πρίστινα. Όπως γνωρίζετε, ο διάλογος έχει ανασταλεί προσωρινός. και γι' αυτό δεν ευθύνεται η Σερβία, αλλά η κυβέρνηση της Πρίστινας, η οποία έχει διαταράξει τη σταθερότητα καθότι εισήγαγε δασμού σε επίπεδο 100% ε, και έτσι παραβίασε τις διευθετήσεις του παρελθόντος με την θέσπιση του λεγόμενου στρατού του Κοσμοπεδίου, με την προσπάθεια ένταξης στην Ίντερπολ χωρίς την Συμφωνία των Βρυξελών και με προκλήσεις κατά της Σερβικής Δημοκρατίας και της ε, Σερβικής ε, Κοινότητας στο Κοσμοπέδιο Μετόχια. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε τέλμα σε ό,τι αφορά αυτό το διάλογο, γιατί η Πρίστινα έχει υιοθετήσει μια θέση διαπραγμάτευσης ε, που ε, απορρίπτει και αρνείται ε, τα επιτεύγματα των διαπραγματεύσεων σε προηγούμενο στάδιο και έτσι έχει ανασταλεί όλη η διαδικασία. Τους προηγούμενους μήνες στο Βελιγράδι μας επισκέφθηκαν εκπρόσωποι της Αμερικανικής Διπλωματίας και ο κύριος Χίλ, καθώς και σύμβουλοι ε, της Άγγελα Μέρκελ ε, και ο Ρίτσαρτ Μούρ από το Υπουργείο Εξωτερικών. Όμως, ε, και πάλι, η Πρίστινα αρνήθηκε να καταργήσει τους δέσμους αυτού, αυτούς. Είναι κρίσιμο σημείο η εξέβρεση ε, ενός κοινού τόπου προκειμένου να συνεχιστεί η ευρύτερη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων. Και πάλι τίθεται θέμα της ασφάλειας της ε, σερβικής κοινότητας στο κοσμοπέδιο και η διασφάλιση ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς μας ε, στο κοσμοπέδιο και τη μετόχεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η κατασταλτική στάση ε, της κυβέρνησης της Πρίστινα και ε, αυτή η, η εθνικιστική ρητορική που ακολουθεί είναι πολύ επικίνδυνη. Η βία που ακολούθησε την σύλληψη του Μάρκο Ντούριτς ε, πέρυσι έδειξε ότι η Πρίστινα είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει βία για να παρεμποδίσει τη διαδικασία. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου μας, του κ. Αλεξάνδρου Βούτσιτς, πέρσι το Σεπτέμβριο και κατά την ε, βίαιη εισβολή ορισμένων μονάδων στο κοσμοπέδιο. Η κατάσταση επιτόπου λοιπόν έχει ε, γίνει πολύ πιο δύσκολη και η Πρίστινα αντιστέκεται σε οποιαδήποτε έστω και περιορισμένη πρόοδο είχαμε επιτύχει. Δεν ακολουθεί τις δεσμεύσεις και τις προθεσμίες που προκύπτουν από τη συμφωνία της 25ης Ιουλίου του 2015. Η Σερβία θα συνεχίσει να διαδραματίζει επικοδομητικό ρόλο για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ένταξης και ολοκλήρωσης θα πρέπει να προωθεί πιο στενή συνεργασία και να αποτρέπει την οικονομική και πολιτική αστάθεια. Γι' αυτό και περιμένουμε να τύχει δίκαιης μεταχείρισης ε, το Βελιγράδι σε ό,τι αφορά τις ε, προενταξιακές διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω σε περιπτώσεις όπου άλλοι φορεί της περιοχής δεν δείχνουν την αντίστοιχη υπευθυνότητα που δείχνουμε εμείς για τη σταθερότητα στην περιοχή. Το κράτος δικαίου σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση και φαντάζομαι γνωρίζετε τι έχει γίνει τελευταία, σε σχέση με την συνταγματική αναθεώρηση και τις σχετικές τροπολογίες. Βλέπουμε ότι η Σερβία δείχνει μεγάλο σεβασμό σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του συστήματος δικαιοσύνης, το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το Μάιο του 2017 η Σερβική Δημοκρατία ξεκίνησε μία ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος δικαιοσύνης ε, και οι συνταγματικές τροποποιήσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτής της γενικότερης μεταρρύθμισης. Έγιναν έξι γύρι στρογγυλής τραπέζης, καθώς και δημόσιος διάλογος στον τομέα των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων και με εκπροσώπους φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Η διαδικασία αυτή ήταν διαφανής και συμπεριληπτική. Ο δημόσιος διάλογος για τις ε, συνταγματικές ε, μεταρρυθμίσεις συνεχίστηκε το 2018 μετά τη δημοσίευση του προσχεδίου στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή της Βενετίας, είναι σημαντικό να το επισημάνω, ε, επισκέφθηκε το Βελιγράδι το Μάιο του 2018. και στην 115η Ολομέλεια ε, ενέκρινε την υιοθέτηση των ε, τροπολογιών. Τον Οκτώβριο του 2018 η Επιτροπή της ε, Βενετίας ενημερώθηκε και παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος και η γνωμοδότηση που εξέδωσε ήταν ότι η αναθεώρηση αυτή συνάδει με τις ε, συστάσεις της. Το Νοέμβριο του 2018 η Σερβική κυβέρνηση υιοθέτησε τις ε, προτινόμενες τροποποιήσεις προς το Σύνταγμα και τις προώθησε στην ε, Εθνοσυνέλευση σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση στα μέσα ενημέρωσης. Το Νοέμβριο του 2017 έγινε μια ειδική συνάντηση με την Ένωση των Δημοσιογράφων που εκδήλωσαν τη δυσαρέσκειά τους προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα και να ε, βρουν ορισμένες λύσεις. Πρότειναν ένα συγκεκριμένο θεματολόγιο ως ε, προαπαιτούμενο Λοιπόν, ήταν η συμμετοχή τους ε, στη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής για τα μέσα ενημέρωσης. Και υπήρξε και μία συνολική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάιο σχετικά με την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης. Από την έκθεση αυτή λοιπόν προκύπτει ότι η κυβέρνηση καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ό,τι αφορά την εφαρμογή του νόμου για την βελτίωση της κατάστασης ε, στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, Ο κερδοσκοπικός ανταγωνισμός έχει οδηγήσει σε ε, υπονόμευση του συστήματος ε, υποβολής ε, εκθέσεων. Τον ε, περσινό Ιούνιο, λοιπόν, ξεκίνησε μια διαδικασία αναθεώρησης του συστήματος με ένα ειδικό σώμα συνεργασίας με τα μέσα ενημέρωσης που θα πρέπει να συνεργαστεί με ομάδα ε, που, στην οποία θα εκπροσωπούνται τα μέσα ενημέρωση για την βελτίωση των σχέσεων και την επίλυση των ανοιχτών θεμάτων. Τον προηγούμενο μήνα έλαβε χώρα και μία δημόσια συζήτηση για την προτινόμενη στρατηγική για τα μέσα και Μέχρι τα τέλη Απριλίου αναμένεται να υιοθετηθεί η νέα στρατηγική και κατόπιν θα τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία. Τώρα, για την ε, πρόληψη της διαφθοράς. Μετά τον διορισμό νέου διευθυντή του Οργανισμού Καταπολέμησης της Διαφθοράς, στα τέλη του 2017, Συνεχίζεται η προσπάθεια για την ε, υιοθέτηση νέου νομοσχεδίου. Υπήρξε και η διαδικασία αδελφοποίησης με Ιταλικές και Ισπανικές αρχές στο πλαίσιο της καταπολέμησης διαφθοράς. Ξεκίνησε η διαδικασία το 2016 και έληξε τον Ιανουάριο του 2019. και αυτό μας βοήθησε πολύ να συντάξουμε τις ε, αλλαγές στο νομικό πλαίσιο. Only few, few, few more sentences and I will finish. Let's go. Επανέρχομαι λοιπόν νομοσχέδιο για την πάταξη τη διαφθοράς. 10 Ιουλίου 18 θα υποβληθεί το σχέδιο. Εν τω μεταξύ εστάλησαν διάφορα άλλα έγγραφα τον Αύγουστο του 18 στην Κομισιόν και η Κομισιόν απήντησε είπε ότι πρέπει να επισκεφθεί η χώρα η Επιτροπή Γκρέκο, πράγμα το οποίο έγινε και αφού ελήφθη υπόψη η άποψη, οι απόψεις των μελών της Γκρέκο το τροποποιημένο νομοσχέδιο υποφλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση φέτος 15 Μαρτίου. Ελπίζουμε ότι η δημοσία συζήτηση επί του νομοσχεδίου θα αποτελέσει μια διαδικασία διαφανή, χωρίς αποκλεισμού και έτσι θα καταλήξουμε σε ένα νέο σύνολο κανόνων όσον αφορά το νέο αυτό όργανο πάταξης της διαφθοράς. Αυτός ο οργανισμός ε, θα έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ε, συγγνώμη που επεκτάθηκα σε λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι αυτές οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Μιλέτσιτς. Στην αρχή είπατε ότι θα είστε σύντομο. Ήμουν αισιόδοξο, η αισιοδοξία μου όμως αυτή ήταν βάσιμη τελικώς. Και δεν θέλω να με παρεξηγήσετε. Έχουμε 11 ακόμη μιλητές. Και έτσι ο χρόνο που απομένει για καθέναν από αυτού θα είναι λιγότερο εξαιτία τη δική σα παρέμβαση. Λυπούμε πολύ, λέει ο ε, Εξαιρετική παρουσίαση, αλλά ζούμε στην πραγματική <laughs> πραγματικότητα και ο, ο χρόνο είναι πάντα εχθρό. Έχουμε ακόμα 34 λεπτά μόνο για αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη κυρίες και κύριοι. Οπότε, τώρα, ο κύριο ε, Τσάμπα, ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ρουμανίας, που ασκεί και την ε, εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Κούτσεν. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Είμαστε όντως από τους λίγους που δεν ήξεραν για την αξία της ένταξης και ξέρω και τι ε, διεργασίε που θα οδηγούσαν προς ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Τελικά καταλήξαμε με τη Λισαβόνα. Λοιπόν, ε, συμπρόεδροι κύριε και κύριοι, εκ μέρου της Προεδρίας του Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην 10η Σύνοδο της ε, Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης και Σταθεροποίησης. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Προεδρίας. Η συνοδο της Διακοινοβουλευτική επιτροπης συνδεσης και σταθεροποίηση. σας μεταφερω τους χαιρετισμού τη Προεδρία. η ρουμανια η Βουλγαρία και η Ελλάδα αξιοποίησαν τις τετραμερείς για να προωθήσουν την την υποψηφιότητα της Σερβίας. Θα έχουμε σύντομα και άλλη μια ε, τετραμερή Βουλγαρίας, Ελλάδας, Σερβίας. Σερβίας και Ρουμανίας. Και τούτο διότι θέλουμε να προωθήσουμε την σταθερότητα και την ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια, στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας. Η ευρωπαϊκή προοπτική πρέπει να ενισχυθεί βάσει της πρόοδου που θα σημειώσει κάθε χώρα και της στήριξη των κριτηρίων. Πρόκειται για την πολιτική διεύρυνση που προωθείται με τι σχετικέ συμφωνίε και τι αποφάσει του Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα, τη Ρουμανία, προσβλέπουμε στο ετήσιο ανακοινωθέν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα μας ενημερώσει για το που βρίσκονται ακριβώς οι, διε... οι μεταρρυθμίσεις στην Σερβία και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Πιστεύουμε ότι ο διάλογος ε, στα Δυτικά Βαλκάνια, θα βοηθήσει την επίτευξη των στόχων της διεύρυνσης. Η διαδικασία Ελιζέ μας εμπνέει και αυτή, καθώς και το γαλλογερμανικό σύμφωνο φιλίες. Αυτά μπορούν να γίνουν και στα Δυτικά Βαλκάνια, ώστε να αφήσουμε επιτέλους την ιστορία πίσω μας. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω περισσότερης εκπαίδευσης για τους λόγους της περιοχής. Επίσης, οι νέοι της περιοχής έχουν ευρωπαϊκές βλέψεις. Το Βουκουρέστι έχουμε μια σχετική σύνοδο. Θα υποστηρίζουμε φυσικά την προοπτική της Σερβίας. Θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τις συνομιλίες. Γίνονται πολλά προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζουμε ότι θα ανοίξουν και περισσότερα κεφάλαια τον Ιούνιο. Θα υπενθυμίσω ότι η πρόοδος εξαρτάται από την πρόοδο που θα σημειώσει η Σερβία εσωτερικά και χρειάζονται περισσότερε προσθέσει, ειδικά στον τομέα του κράτου δικαίου. Είμαι την ευκαιρία να συζητήσουμε στο Βουκουρέστι με όλε τι υποψήφιε χώρε και στο πλαίσιο τη άτυπη υπουργική. Είχαμε και συνάντηση με του επικεφαλεί των αντιπραγματεύσεων με όλε τι υποψήφιε χώρε. Εκεί συζητήσαμε, προέβημε σε επισκόπηση τη πρόοδου σε όλε τι χώρε, με ιδιαίτερη όμω έφαση στην Σερβία τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η οικονομική διακυβέρνηση, όλα αυτά παραμένουν τα κυριότερα ζητήματα στην διαδικασία ένταξης. Αυτό υπεγράφει και στην τελευταία σύνοδο 18 Δεκεμβρίου που είχαμε με την Σερβία και καλέσαμε την Σερβία να λάβει υπόψη της, τα συμπεράσματα και τι συστάσει να βελτιώσει τι επιδόσει τη στην δημοκρατική διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, την ελευθερία τη έκφραση των μέσων, την πάταξη τη διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματο. Η υλοποίηση στα κεφάλαια 23 και 24 παραμένει βασική σημασία. Πρέπει να ληφθούν λοιπόν οι υπόψη πρόοδος στην επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων. Όλα αυτά θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο, όπως επίσης ρόλο θα παίξει και η επιχείρηση των μειονοτήτων. Εδώ η κυβέρνηση της Σερβίας νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά, πρέπει να κάνει πολλά, να κάνει κινήσεις ε, που θα μεταφραστούν και σε νομοθεσία. Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης την ελευθερία της εκφράσης των μέσων, την προστασία της ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Αναγνωρίζουμε τις πρωτοβουλίες Προέδρου και Πρωθυπουργού να ξαναγράψουν τη σχετική νομοθεσία χωρίς αποκλεισμούς με τρόπο αυτοσυνεπή. Υπενθυμίζουμε τι δεν πάει καλά στην ελευθερία της έκφρασης. Τα προβλήματα αυτά είναι απόλυτης προτεραιότητας. Οικονομική διακυβέρνηση και εδώ έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις στην Σερβία. Έχουμε καλή πορεία της σερβικής οικονομίας, σταθεροποίηση των τιμών και του πληθωρισμού, καλές γενικές επιδόσεις, αλλά και εδώ Χρειάζεται κάτι περισσότερο για να συνεχιστεί η ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε περισσότερες μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς και δημοσιονομική πειθαρχία. Συγχαίρουμε επίσης την Σερβία για τις προσπάθειες στην πάταξη των ε, παρατυπών μεταναστευτικών ροών. Έχουμε καλύτερη διαχείριση των συνόρων, καλύτερη συνεργασία με τους γείτονες, πάταξη του λαθρεμπορίου. Και με την ευκαιρία υπενθυμίζω ότι ως υποψήφια χώρα η Σερβία πρέπει να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους τομείς. Στις προσπάθειες, για παράδειγμα, ακολούθηση της ε, ΚΕΠΑ και ΠΑΑΜ και η Σερβία μπορεί να κάνει περισσότερα. Η έλλειψη ευθυγράμμισης κάποιες ε, αποκλήσει ε, σε επίπεδο πολιτικής αποτελεί πηγή ανησυχία. Η καλή πολιτική γειτονία είναι κομμάτι τη ένταξη βεβαίω. ξέρουμε ότι η Σερβία έχει λάβει επικοδομητικά μέτρα στην περιοχή αυτή του κόσμου. Χρειάζεται όμω περισσότερη πρόοδο στι σχέσει καλή γειτονία και διαχείριση των συνόρων. Και όλα αυτά σε συμφωνία βεβαίω με το διεθνέ δίκαιο. Όσον αφορά την εξομαλύνση των σχέσεων με την Πρίστινα, σίγουρα μπορούν να αξιοποιηθούν εδώ ε, η βοήθεια μεταξύ άλλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβουλίο θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα εν ώψη της συνέχισης των διαπραγματεύσεων επί του κεφαλαίου 35. Οπότε κυρίε και κύριοι, να πω κατακλείδη ότι πρέπει να αξιοποιήσει η Σερβία τις καλές συνθήκες αυτή τη στιγμή, να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να ενημερώσει τον πληθυσμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικό εταίρο τη Σερβία σε όλου του τομεί και πρέπει την στρατηγική αυτή επιλογή να τη στηρίξει η Σερβία δημοσίω. Συγχαρητήρια επίση για την προσήλωση τη εργασία αυτή τη Επιτροπή. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σα στην πρόθεση των σχέσεών μα. Εκτιμούμε βαθύτατα και την υποστήριξη συναφώς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την υποστήριξή σας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Μακρύβης, αναπληρωτής επικεφαλής ε, του Τμήματος Σερβίας. Πρόεδρε, κύριε, συμπρόεδροι, κύριε και κύριοι, θα προσπαθήσω να είμαι ακόμα πιο σύντομος από ό,τι θα ήμουν. να πω πρώτα απ' όλα ότι το 2018 ήταν ένα σημαντικό έτος το οποίο εμπέδωσε τις σχέσεις της Σερβίας με τα Δυτικά Βαλκάνια. Τον Φεβρουάριο είχαμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής από την Κομισιόν. Τον Μάιο είχαμε την σύνοδο στη Σόφια και τη σχετική δήλωση καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ελπίζουμε ότι το 2019 θα συνεχίσει να εξελίσσεται προς την ίδια κατεύθυνση και θα ενισχύσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή πρόπτικη των Δυτικών Βαλκανίων. Πολύ σύντομα στο Βελιγράδι θα έχουμε την ψηφιακή σύνοδο των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για το Βελιγράδι να διδραματίσει σχετικό ρόλο στην υλοποίηση της ψηφιακής θεματικής στα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης, αυτό είναι ένα καλό βήμα και για την έκτη σύνοδο Βερολίνου στο Κώστεν, οι διαπραγματεύσει με την Σερβία ήδη αναλύθηκαν με αρκετέ λεπτομέρειε, οπότε δεν θα επαναλάβω τα όσα ήδη ακούστηκαν. Δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, ο ρυθμό τη εξέλιξη των διαπραγματεύσεων είναι στα χέρια τη Σερβία. Εξαρτώνται δηλαδή από τι μεταρρυθμίσει τη Σερβία σε όλου του τομεί και δι στο κράτο δικαίου και στην εξομάλυνση των σχέσεων με το Κωσυφοπαίδιο. Αυτά λοιπόν θα καθορίσουν την ταχύτητα των διαπραγματεύσεων. Δεύτερον, όπως ακούσατε και από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κύριο έχουμε και θέματα τα οποία μπορεί να είναι αόρατα ούτως όμως πρόκειται για θέματα από των οποίων έχουμε μια σιωπηρή συνεργασία με την κυβέρνηση και κάθε φορά που έχουμε ένα κείμενο από την κυβέρνηση να ξέρετε ότι αυτό σημαίνει ότι έχει επιτελεστεί πολύ σημαντική πρόοδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι πολύ καλό, είναι καλό σημάδι και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία και σε αυτού του τομεί. Δύο πράγματα για την υποστήριξη που συζήτησαμε προηγουμένω από την πλευρά της Κομισιόν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την Σερβία στον δρόμο της προς την Ευρώπη. Όπως προείπαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος, υπερθούν ένα στρατηγικός και οικονομικός εταίρος. Είναι ο μεγαλύτερος δωρητής. Δεν υπάρχει σύγκριση με κανέναν άλλον εταίρο της Σερβίας. Το Υπουργείο Ευρωπαϊκή Πολιτικής διενεργεί διάφορε δημοσκοπήσει. Η τελευταία έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο. Και τον Δεκέμβριο ήταν και η πρώτη φορά που οι Σέρβοι αναγνώρισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον μεγαλύτερο δωρητή, μεγαλύτερο από την Ρωσία. Αυτό είναι θετική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, η τάση είναι άλλη. Δηλαδή, τα αποτελέσματα τη δημοσκόπηση δεν αποτυπώνουν το μέγεθος της οικονομικής βοήθειας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αξίζουμε αναγνώρισης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στο πλαίσιο της στρατηγικής δέσμευσης της χώρας στον δρόμο της ένταξης. Τα νούμερα είναι αδιάψευστα. Τα τελευταία δέκα χρόνια η Σερβία έλαβε πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ δωρεάν επιχορηγήσεις. Μιλάμε για κονδύλια τα οποία δεν επιστρέφονται είναι δώρο προς τη χώρα. Ας δούμε όμως και το εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το εμπόριο είναι μια συμπαγής ιδιαίτερο συμπαγή οντότητα, δύο τρίτα του εμπορίου τη Σερβία διεξάγεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη θέση σε ισχύ τη Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση το 2008, οι εξαγωγέ τη Σερβία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση τριπλασιάστηκαν. Πρόκειται για εξαγωγές που αυξάνονται κάθε χρόνο κατά 10%. Άμεσες ξένες επενδύσεις. Η Σερβία είναι πλέον ένας πολύ ελκυστικός προορισμός για ευρωπαϊκές επενδύσεις. 73%. Το παραλαμβάνω. 73% των ξένων αμέσων επενδύσεων στην Σερβία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ 2010 και 2017, σωρευτικά, οι εισρωές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται σε 11,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η υποστήριξη αυτή είναι και η καρδιά του ζητήματος. Αυτά ξέρετε ενδιαφέρουν τους Σέρβους. Ενδιαφέρουν την οικονομία, την ευμερία, την κοινωνία των πολιτών, το κράτος δικαίου. Εκεί έγκυται η ουσία των σχέσεών μας. Είμαστε κοντά στην Σερβία, να ξέρετε, και η προοπτική ένταξη της Σερβία μας φέρνει ακόμη πιο κοντά. Και τώρα δύο άλλες πτυχές της διαδικασίας ένταξης που είναι σημαντικές και που καθορίζουν την ταχύτητα των διαπραγματεύσεων. Πρώτον, δημοκρατική διακυβέρνηση κάτι το οποίο πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα για την Σερβία. Προκειμένου ο ρόλο του Κοινοβουλίου, πρόθεση δηλαδή τη θεματική της Ευρωπαϊκή Ένωση, η λογοδοσία τη κυβέρνηση, εδώ όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι διαδικασίε που παρακολουθούμε, πρόκειται για νομοσχέδια που πρέπει να εγκριθούν τάχιστα στην Σερβική Βουλή. Δυστυχώ το έργο του Κοινοβουλίου, το νομοθετικό αλλά και το ελεγκτικό, δεν έχουν πάει καλά τα τελευταία, του τελευταίου μήνε με αποτέλεσμα νομοσχέδια όπως ο προπολογισμό του 2019 δεν προχώρησαν. Η χρήση της κατεπίγουσας διαδικασίας ε, έχει γίνει αντικείμενο κατάχρησης. Χρειάζεται λοιπόν πιο ποιοτικό πολιτικό διάλογο για να λειτουργήσουν πραγματικά οι δημοκρατικοί θεσμοί στη Σερβία. Πιστεύουμε ότι ο πολιτικό διάλογο πρέπει να παραμείνει εκεί που ανήκει, δηλαδή στη Βουλή ο δημοκρατικός χώρος για την αντιπολίτευση εντός της Βουλής πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από Σε αυτό είναι κατεπήγον θέμα, είναι κατεπήγουσα ανάγκη και αυτά πρέπει να γίνουν, επαναλαμβάνω, εντός της Βουλής, εντός του Σερβικού Κοινοβουλίου. Τέλος, να πω αυτό που είπαν και οι ευρωβουλευτές στο Βελιγράδι, το είπε και ο κύριος Κούκαν λίγο πριν. Έχουμε και τον διάλογο Ζαν Μονέ. Τον υποστηρίζουμε, Ελπίζουμε ότι θα αξιοποιήσετε αυτήν την δυνατότητα εσείς οι συνάδελφοι από την Σερβία. Και για να έρθουμε στο κράτος δικαίου, δύο πτυχές του θέματος. Το πρώτο είναι η δικαιοσύνη. Οι τροποποιήσεις του συντάγματος πρέπει επιτέλους να εγκριθούν και να υλοποιηθούν. αλλά χρειάζονται και άλλα νομοσχέδια και όλα αυτά με τρόπο, όπως είπα, χωρίς αποκλεισμού με διαφάνεια και σε συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας. Ελευθερία της έκφρασης. Και εδώ θέλουμε να δούμε περισσότερη πρόοδο. Τα καλά νέα όμως είναι ότι έχουμε μια νέα στρατηγική για τα μέσα, για τα ΜΜΕ. Άνοιξε μια ματιά στους στόχους της νέας στρατηγικής ε, διαπιστώσετε ότι για πρώτη μάλλον φορά συμφωνούμε ως προς τις διαπιστώσεις με τις σερβικές αρχές. Το σχέδιο αυτό στρατηγικής είναι κατηγορηματικός προς τις ε, επιθέσεις κατά των δημοσιογράφων όσον αφορά την διαφάνεια και όσον αφορά την συγχρηματοδότηση από δημόσιους φορείς με σκοπό την εξασφάλιση ανεξαρτησίας στα κρατικά μέσα. Τώρα, εν ώψη τη ε, υλοποίησης, έγκρισης και υλοποίησης της στρατηγικής. Ε, αυτά είναι τα σημαντικά γιατί τελικώ ε, καλή θεωρία, αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να τα δούμε όλα αυτά εφαρμοσμένα στην πράξη. Οικονομία. Συζητήσαμε πολλά. Συγχαρητήρια στην Σερβία για την πρόοδό τη. Ενθαρρύνουμε την Σερβία να συνεχίσει τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων για να μπορέσει ακριβώς να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες. Οπότε κλείνω εδώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματο τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, ο κύριο Ραμπόν. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη, είναι μεγάλη τιμή για μένα που παίρνω τον λόγο να πιάσω σήμερα. Θα είμαι σύντομο, ε, κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε ότι Υπάρχει μεγάλη προσήλωση και σημαντικές εξελίξεις. Είχαμε την ομιλία ε, του κ. Γιούνκερ το 2017, τον, ε, τη για τα Δυτικά Βαλκάνια επίσης το 2017, τα συμπέρασματα του Συμβουλίου μετά τη, και μετά τη Σύνοδο του Λονδίνου. Αυτό δείχνει ότι όλη η περιοχή μαζί με τη Σερβία είναι σημαντική και αυτό δείχνει πόσο σημαντικά εξετάζουμε την πρόοδο των ε, προεντεξιακών διαπραγματεύσεων. Τώρα έχει έρθει η ώρα να δούμε πώς μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δεδομένου ότι και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι προτεραιότητα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του, της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για να γίνει αυτό πρέπει βέβαια η Σερβία να μας δώσει τα απαραίτητα αποτελέσματα ε, στη μεταρρύθμιση, στο κράτος δικαίου, στο σύστημα δικαιοσύνης, στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερία του τύπου. Αντίστοιχη πρόταση θα πρέπει να σημειωθεί και στην εξομάλυνση στο σχέση με, την, ε, με το κοσμοπέδιο. Όλα αυτά είναι πολύ κρίσιμα για την πρόοδο των πρωτεξιακών διαπραγματεύσεων. Το δικαίωμα στι ειρηνικέ διαδηλώσει είναι βασικό στοιχείο και θεμελιώδη αξία τη δημοκρατία και θα πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστή. Οι διαδηλώσει λοιπόν θα πρέπει να γίνονται ειρηνικά και σύμφωνα με τον νόμο. Με και φυσικά ο πολιτικός διάλογος ε, θα πρέπει να διεξάγεται στο Κοινοβούλιο. Αντίστοιχα, το δημοκρατικό περιθώριο ε, και για την αντιπολίτευση εντός του Κοινοβουλίου θα πρέπει να διασφαλίζεται. Τον τελευταίο χρόνο είδαμε ότι υπήρχε έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου σε σημαντικές νομοθετικές προτάσεις. Σε ό,τι αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και άμυνας, υπάρχει έντονη συνεργασία με τη Σερβία. Συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στις ε, αποστολές και επιχειρήσεις μας, σε τέσσερις ε, στην Αφρική, στο Μαλί, στην ε, Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, στη Σομαλία. Το Βελιγράδι τώρα προετοιμάζει το πλαίσιο για να συμβάλλει και σε μη στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι η πρώτη χώρα αυτής τη περιοχής ε, που συμβάλλει με τέτοιο τρόπο. Συμμετέχει και ε, στην ομάδα κρούση EU Hellbrook και σε άλλα προγράμματα. Ταυτόχρονα όμω ε, δεν ευθυγραμμίζεται με μια σειρά θέσεων σε ό,τι αφορά την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλεια. Και υπάρχει υπαναχώρηση τα τελευταία χρόνια υπογραμμίζουμε εκ νέου την έκκλησή μας προς Σερβία να συνεχίζει να ευθυγραμμίζεται με την κοινή εξωτερική ε, πολιτική πολιτική ασφαλείας. Είχαμε και την τελευταία τέτοια συνεδρίαση στις Βρυξέλλες πέρυσι. Υπάρχει σαφή σχέση ε, μεταξύ της υιοθέτησης αυτών των στόχων και της πρωτεξιακής πορείας της χώρας. Αυτό επισημάνθηκε στην ε, τελευταία συνάντηση. Η ανάγκη για το Κοσμοπέδιο και τη Σερβία να διασφαλίσουν ένα διάλογο, ένα πλαίσιο που ε, προωθεί και επιτρέπει αυτόν τον διάλογο, προκειμένου να υπάρχει εξομάλυση των σχέσεων. Οι δεσμοί που έχει επιβάλει το Κοσμοπέδιο θα πρέπει να καταργηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ράμπολτ. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα η κυρία Κόβατς. Μετά ο κύριος Μακάλιστερ. Στην πρώτη μιλήτρα να πω ότι αν τηρήσεις ε, το πεντάλεπτο θα σου πάρω παγωτό. Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να μείνω και κάτω από τα 5 λεπτά. Γιατί έχει και ωραίο καιρό έξω και θα το ήθελα αυτό το παγωτό που προτείνατε. Η Σερβία φυσικά έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσει ε, να πληρεί τις προϋποθέσεις. Έχουμε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ε, πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία, καθότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί η αξιοπιστία μας. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε την ε, ευρωπαϊκή μας προοπτική, αυτή η στήριξη να είναι σταθερή και ανυποχώρητη. για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό προκειμένου να συνεχίσουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις που πετούνται για να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το άνοιγμα των κεφαλαίων, αλλάξαμε το νομικό μας πλαίσιο, υιοθετήσαμε μεταρρυθμίσεις, αλλάζει και η κοινωνία μας. Ακόμα και τώρα που βρισκόμαστε στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καταληκτική προθεσμία για αυτές τις πραγματεύσεις και τα πάντα εξαρτώνται από την ε, πρόοδο που σημειώνουμε. Και δυστυχώς δεν μας ικανοποιεί ο αριθμός των ε, κεφαλαίων που έχουν ανοίξει μέχρι τώρα. Υπάρχουν πολλές ε, υποχρεώσεις και από πλευρά θεσμικών οργάνων στη Σερβία με πολύ σημαντικές προκλήσεις για την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό ολόκληρη κοινωνία να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά για τη Σερβία η στόχη είναι σαφής. Θέλουμε να γίνουμε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πλευράς μας το σημαντικό είναι οι μεταρρυθμίσεις ε, να ανήκουν εντό αγωγικών στην υποψήφια χώρα η ποιότητα των διαπραγματεύσεων είναι πολύ πιο σημαντική από τον αριθμό των κεφαλαίων που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Ο αριθμός των ανοιχτών κεφαλαίων δεν αποτελούν ε, ε, ακριβές κριτήριο του συνόλου της διαδικασίας. Το σημαντικό είναι να επενδύσουμε στην ευημερία, τη δημοκρατία, τη σταθερότητα ολόκληρης της ε, Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ακούσαμε και τον συνάδελφο Όρλιτς προηγουμένως. Ε, πράγματι, είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στους πολίτες μας τα ωφέλη της ε, ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό με ακόμα πιο δραστήριο τρόπο, να υπάρξει σωστή επικοινωνία αυτού του μηνύματο. Υπάρχει όμως πολύ σημαντικός αριθμός ε, Σέρβων πολιτών που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή μας προοπτική. Και την τελευταία δημοσκόπηση φάνηκε ότι η νέα μας στρατηγική προβολή των ευρωπαϊκών δωρεών αποφέρει καρπούς. Βλέπουν λοιπόν και αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι Σέρβοι πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο υπαριθμόν ένα ε, δωρητής στη Σερβία. Οι πολίτες μας είναι σημαντικό να δουν και όλα τα ωφέλη να δουν ότι βελτιώνεται το βιωτικό τους επίπεδο, η καθημερινότητά τους. Ξέρουμε ότι η διπραγμάτευση δεν προχωρεί αυτόματα. Πρέπει και εμείς ε, να πετύχουμε τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται. Και από εκεί θα εξαρτηθεί και ο δρόμος μας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστρέφω τώρα λοιπόν στα κεφάλαια. Για να είμαστε ειλικρινοί, στα τελευταία πέντε χρόνια η Σερβία διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει ανοίξει όμως ε, το 50% των κεφαλαίων και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το άνοιγμα των κεφαλαίων προς διαπραγμάτευση ε, ξέρουμε ότι δεν είναι τίποτα μπροστά στο κλείσιμο των ε, κεφαλαίων. Πολύ δουλειά λοιπόν απομένει. Κάθε εξάμεινο η Σερβία ανοίγει δύο κεφάλαια, ενώ κανονικά θα πρέπει να ανοίγει πολύ περισσότερα. Και αυτό ισχύει εδώ για πολλά χρόνια. Μου λένε λοιπόν πρέπει να κλείσω σιγά σιγά. Θεωρώ ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου και ο ρόλος ε, αυτής της Επιτροπής είναι να εξεκολουθεί να εργάζεται προς την υιοθέτηση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων με βάση τον τελικό μας ε, στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Κοντά ήσασταν, αλλά όχι ακριβώς στο πεντάλεπτο. Το λόγο έχει τώρα ο Ντέιβιτ Μακάλιστερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων και μόνιμος ε, εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Σερβία. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ, Edward. Μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Αγαπητοί φίλοι από τη Σερβία, αγαπητοί συνάδελφοι. Πέντε παρατηρήσεις από πλευράς μου. Πρώτον, η Σερβία βρίσκεται στο δρόμο προς την ευρωπαϊκή ένταξη. Δεν έχει να κάνει με τις προθεσμίες και τις ημερομηνίε, έχει να κάνει με τα αποτελέσματα. Συνεχίστε λοιπόν τη σκληρή δουλειά που κάνετε αυτή τη στιγμή για να βελτιώσετε και την απόδοσή σας. Δεύτερον, το κράτος δικαίου, όπως ακούσαμε και πάλι σήμερα, βρίσκεται στο επίκεντρο των ε, προενταξιακών διαπραγματεύσεων. Τρίτον, η ελευθερία του τύπου των μέσων ενημέρωση θα πρέπει να ε, είναι δεδομένη, είναι κάτι το θεμελιώδες ε, για μια δημοκρατία. Πρέπει να προχωρήσετε στην πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών στις οποίες έχετε καταλήξει, να συνεχιστεί ο διάλογος με την Πρίστινα και πέμπτον να ενισχύσετε τον ρόλο του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τη ε, συζήτηση και εξέταση της νομοθεσίας. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουν πει οι προηγούμενοι μιλητές. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, Σέρβους φίλους μας που ταξίδεψαν μέχρι το Στρασβούργο και πάλι για μια τελευταία φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας και να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και τον ε, συμπρόεδρο Βλάντιμιρ Όλιτς για την πολύ καλή συνεργασία με μένα ως εισηγητή και κλείνοντας να ευχαριστήσω και τον αξιότιμο συνάδελφο Edward Κούκαν. Όπως ξέρετε δεν θα θέσει ξανά ψηφιότητα στις επερχόμενες ευρωεκλογέ. Και μια προσωπική παρατήρηση. Σας ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιάς για το πολύτιμο έργο σας. Ε, θα μας λείψετε πραγματικά. Έχετε αποδείξει ότι είστε πραγματικός φίλος της Σερβίας. Ευχαριστώ. Θα σε κεράσουν δύο μπύρες μετά. σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα να συνεργαστώ μαζί σας. Ο κύριος Σόρμας έχει το λόγο τώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Υπάρχουν ορισμένα σημεία και ζητήματα που ανακύπτουν ξανά και ξανά. Φυσικά και η Σερβία θέλει να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια, οπότε είναι ε, δεδομένο και αυτονόητο ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα δικαιοσύνη μας. Όλα αυτά τα, έχετε, τα έχουν ήδη θίξει οι προηγούμενοι μιλητές. Όλα αυτά μπορεί να επιτευχθούν όμως πολύ πιο εύκολα Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε ένα κεφάλαιο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ανοίγουμε περισσότερα κεφάλαια. Κεφάλαια που είναι έτοιμα να ανοιχθούν. Ακούσατε ότι υπάρχουν πέντε τέτοια κεφάλαια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ανοίγουν. Γιατί ακόμα και αν ανοίξουμε αυτά τα κεφάλαια, δεν σημαίνει ότι θα μπει αυτομάτω η Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώ σημαίνει ότι καθυστερούμε στο έργο μα, ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση τη Σερβική με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι καλύτερο να ανοίξουμε περισσότερα κεφάλαια παρά να αρχίσουμε να κλείνουμε τα υπόλοιπα. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Ο Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στην αρχή της χρονιάς έδωσε έτσι μία επισκόπηση των ε, συστημάτων υγείας ανά την Ευρώπη. Εκεί λοιπόν βλέπουμε. Και εγώ να σας πω φυσικά ότι θεωρώ ότι πρέπει να βελτιωθεί το σύστημά μας. Παρ' όλα αυτά, το σύστημά μας έλαβε καλύτερη αξιολόγηση από 14 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά το σύστημα κατάρτισης, ε, βρισκόμαστε στην τέταρτη θέση. Ή σε ό,τι αφορά την απασχόληση στο μέτρο της πληροφορικής, είμαστε πολύ ψηλά και εκεί. Αυτό σημαίνει ότι η ηγετική θέση η Σερβία, όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην Ευρώπη. Και εγώ βέβαια δεν δηλώνω ικανοποιημένο ε, με τα πάντα. Εγώ είμαι βουλευτής από το 2000. Ε, ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο και ξέρω ότι μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Πρέπει λοιπόν στην Σερβία να εργαστούμε για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντικό να ανοίξουμε περισσότερα κεφάλαια. Όχι για να μπούμε πιο γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να αρχίσουμε αυτή την προσπάθεια, τη διαδικασία εναρμόνισης της νομοθεσίας μας. Έτσι κι αλλιώς, ε, τα πιο σημαντικά επιτεύγματα προκύπτουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε ότι πέρυσι οι επενδύσεις στη Σερβία ε, είναι παραπάνω από τις επενδύσεις ε, στο σύνολο των υπολείπων βαλκανικών χωρών. Φαίνεται λοιπόν ότι Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στη Σερβία και περιμένουμε να έχουμε πολύ μεγάλη επένδυση αυτή τη στιγμή στη Σερβία με την άφηξη της Volkswagen. Α, και ο συνάδελφος ε, σχολιάζει. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και ελπίζω έτσι να καταφέρουμε να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, που είναι ο στρατηγικός μας στόχος ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ντέλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όταν ξεκινήσατε την ομιλή σας, ε, είπατε για νοσταλγία. Όντως πρόκειται για την τελευταία σύνοδο της Επιτροπής μας, Εγώ προσωπικώς είμαι υπερήφανος, φαντάζομαι όλοι μας, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι η αντιπροσωπεία μας, υπό την σας, καθοδηγήσή σας, κύριε Κούκαν, ήταν μία από τους ένας μάλλον από τους στυλοβάτες της διεύρυνσης. Φέτος έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές όπως όλοι γνωρίζουμε, σημαντικές όχι μόνο για το μέλλον εν γέννη, αλλά και για το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων. Τα πέντε προσεχή έτη είναι πολύ σημαντικά για τους δύο πρωτοπόρους, τους δύο προπορευόμενους μάλλον, Σερβία και Μαυροβούνιο. Οπότε μπροστά μα έχουμε πολλή δουλειά για να πετύχουμε του στόχου, το στόχο τη ένταξη και τη διάρκεια τη επόμενη θητεία. Είναι προς το συμφέρον λοιπόν της περιοχής να τύχει ευρεία υποστήριξη και από το επόμενο κοινοβούλιο. Ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι βεβαίω κρίσιμο για άλλη μια φορά. Πάντω, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις σε κρίσιμες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα 100% δασμοί που επέβαλε η Πρίστινα σε σερβικά εμπορεύματα, κάτι το οποίο είναι, σε, είναι αντιδιαμετρικά αντίθετο με αυτό το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να κάνει εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή συνοχή και οικονομική συνεργασία στην περιοχή. Και παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή πάγωσε τον διάλογο μεταξύ των διμερών. Βεβαίω, όπως είπε η κυρία Πρέσβης, και το μάθαμε και από τις δημοσκοπήσεις, οι πολίτες της Σερβίας παραμένουν προσιλωμένοι στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας τους. Πιστεύω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλο αυτό εμείς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις πρέπει να επιταχυνθούν. Η πρόοδος γνωρίζουμε στο κεφάλαιο 23 είναι προϋπόθεση για το άνοιγμα και άλλων κεφαλαίων με τη Σερβία, όμως έτσι όπως έχουν τα πράγματα θα ήταν, άδικο να παραμείνει όμοιρος η Σερβία εξαιτία της αδυναμίας και της Ανυκανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει μονομερεί ενέργειε τη Πρίστινας. Οπότε, κατά τη διάρκεια τη επόμενη θητεία, αν είμαστε εδώ μετά το Μάιο, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, διότι τα Δυτικά Βαλκάνια και δι η Σερβία και το Μαυροβούνιο, οι προπορευόμενοι, πραγματικά έχουν μεγάλη ανάγκη και περιμένουν τη βοήθειά μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαριάνοβιτς. Κούκαν, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα συζητούμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Σερβίας. Νομίζω ότι συζητούμε πια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει σχέση. Το ερώτημα είναι αν η πρόοδος αυτή εξελίσσεται, προοδεύει και προς ποια κατεύθυνση από την ίδρυση την ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καθεστική αλήθεια είναι ότι η οικονομική και άλλη σταθερότητα δεν υπάρχει χωρίς κρατός δικαίου, χωρίς σεβασμό για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Σήμερα μετά πολλά χρόνια φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να μας παραφέρουν στο παρελθόν. Εμείς είμαστε υπέρ της συμμετοχής δημοκρατίας, υπέρ της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, υπέρ των ανεξαρτών αρχών, υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης, υπέρ των κοινωνικών δικαιωμάτων. Δυστυχώς για κάποιους, για κάποιες πολιτικές ελίτ, αυτό δεν είναι πλέον το ιδεώδες. Αυτό συμβαίνει για ορισμένους σήμερα στην Σερβία, αλλά και αλλού. Ξέρετε, μετά από τόσου αιώνε υπάρχουν πολλοί ορισμοί τη δημοκρατία. Ένα ορισμό λέει ότι πρόκειται περί διαδικαστικών κανόνων για να παίρνουμε συλλογικά αποφάσει. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για τι αγρότε δυνάμει που διαβρώνουν την δημοκρατία κλπ. Ε, άλλοι πάλι λένε ότι η δημοκρατία είναι ο μόνος τρόπος άσκησης της εξουσίας. Εγώ θα σας μιλήσω σήμερα για την επιδρομή, την, την επιχείρηση κατά της Βουλής. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, μεταξύ άλλων βεβαίω, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μια Βουλή η οποία θέλει να λειτουργεί, να ε, ψηφίζει νόμους και αν η Βουλή δεν λειτουργεί, οι πολίτες δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν υπάρχει διαφάνεια, έχουμε απλώς διαφθορά. Κύριε Είπατε ότι ανησυχείτε διότι μέρος της αντιπολίτευσης μποϊκοτάρει τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Να σας πω δύο πράγματα ως προς αυτό. Η απόφαση να μποϊκοτάρουμε την ολομέλεια της Βουλής και τη λειτουργία της δεν ήταν ομόφωνη. Αναγκαστήκαμε όμως γιατί μετά από έξι χρόνια τυραννίας της πλειοψηφίας η κατάσταση δεν είναι πλέον ανεκτή φτάσαμε να ζούμε σε ένα αυταρχικό σύστημα υπό τον πλήρη έλεγχο ενός κράτους, ε, υπό ενός ενδρός αρχή. Η ελεγκτική λειτουργία της Βουλής έχει ακυρωθεί ε, και τότε ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις από πολίτες με ε, αιτήματα, με ένα τουλάχιστον από τα αιτήματα, η Βουλή να εκπροσωπεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο όσους ασκούν την εξουσία. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ατμόσφαιρα στην Σερβική Βουλή είναι πολύ διαφορετική από αυτήν εδώ. Να σας δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβετε. Είναι και τμήματα της δήλωσης που υιοθετήσαμε. πέραν των διακηρύξεων, δύο μόνο δημόσιε συνεδριάσεις της Βουλής έγιναν, κάτι λιγότερο από μία το χρόνο. Η Επιτροπή Πολιτισμού δεν εξέλεξε καν επίτροπο υπεύθυνο της ανεξάρτητης αρχής για την ενημέρωση. Επιβάλλεται στα μέσα αυτό λογοκρισία και αυτό είναι αποτέλεσμα πιέσεων. Μεγάλο πρόβλημα ε, το οποίο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι του οι δημοσιογράφοι και τα μέσα. Χρειάζονται συστημική αντιμετώπιση όλα αυτά. Γι' αυτό και καλούμε την κυβέρνηση και τα αρμόδια όργανα να υιοθετήσουν την αρχή της κατάργησης των αποκλεισμών, την προστασία των μέσων και όλα αυτά να εφαρμοστούν στην πράξη και για την ελευθερία τη έκφραση. Πρέπει η ρυθμιστική αρχή για τα ηλεκτρονικά μέσα να λειτουργεί με τρόπο διάφανο. Ο διορισμός των μελών αυτής της ενεξάρτητης αρχής πρέπει επιτέλους να γίνει. Έχουμε καθυστερήσει δύο χρόνια. Πρέπει να εμπεδώσουμε τον δημόσιο διάλογο, να δώσουμε τη μάχη των ψευδοειδήσεων, να αποκραστήσουμε τον επαγγελματισμό των δημοσιογράφων. Το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο είμαι μέλος, δεν έχει αλλάξει τη θέση του όσον αφορά την ένταξη της Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε υπέρ βεβαίω τη ένταξης. Είμαστε υπέρ του ανοίγματο νέων κεφαλαίων, όμως ανησυχούμε. Ανησυχούμε διότι η προοπτική αυτή αποδυναμώνεται Λόγω των ζητημάτων που σας προανέφερα, τα φέρα των αξιών μπαίνουν σε δεύτερη ταχύτητα. Δυστυχώ οι δημοκρατικές δυνάμεις έχουν αποδυναμωθεί σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. Έχουμε ακροδεξιές δυνάμεις, ακροδεξιά κόμματα, ε, δεξιά κόμματα στη χώρα μου, τα οποία ήταν στο περιθώριο στο παρελθόν χάρη στην ευρωπαϊκή πολιτική. Πάντως, συγχαίρουμε την κυβέρνηση για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, Αυτό είναι, αυτές είναι καλοδεχούμενες, όμως υπάρχει και άλλη πτυχή. Δεν πάμε μπροστά μόνο με τα μακροοικονομικά δεδομένα, όταν ξέρουμε ότι 400.000 παιδιά είναι πολύ κοντά στο να ζουν στο όριο της φτώχειας. Πρέπει οι πολίτες της Σερβίας να νιώσουν την οικονομική πρόοδο στην πράξη, να ζήσουν επιτέλους σε μια σταθερή και διαφανή αγορά εργασία, να μειωθούν οι διαφορές, οι διαφορές και οι διακρίσεις, να μειώσουμε την φτώχεια. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Επαναλαμβάνω ότι η αντιπολίτευση θέλει να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή, στην πρόθεση της ευρωπαϊκής πολιτικής Σερβία, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο ισότιμο, με τρόπο δημοκρατικό. Δεν θέλουμε να γίνουμε και πάλι, να μπούμε στο στόχαστρο της κυβέρνησης, ούτε να καταγγελθούμε ως υπεύθυνοι για όλα όπως γινόταν επί Μιλόσεβιτς. Ο αγώνας για την εξουσία δεν γίνεται με ισότιμους κανόνες. Το κόμμα στην εξουσία έχει κατακυριεύσει όλους τους μηχανισμούς. Δημιουργεί λοιπόν μια ατμόσφαιρα που δεν είναι αποτεκτή η διαφορά, Θέλουμε ένα κλίμα το οποίο θα σέβεται τις μειονότητες μεταξύ άλλων χωρίς διακρίσεις. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις ε, επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Θέλουμε να δούμε και εμείς μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική, πιο κοντά στους πολίτες της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να σε ενημερώσω ότι ο επόμενος ομιλητή είναι ο κύριο Χοκμάγερα και με ο κύριο Κολομπιέ για την ε, πρώτο ομιλητή για το θέμα του διαλόγου. Όμω, πέντε η ώρα ξέρετε ότι πρέπει να πάμε στην Ολομέλεια γιατί έχουμε ψηφοφορίε. Γκούναρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους Σέρβους συναδέλφους που ήρθαν στο Στρασβούργο. Για μερικούς από εμά είναι δύσκολο λόγω απόσταση, πόσο μάλλον για εσάς. Εγώ είμαι μεταξύ αυτών που ελπίζουν και προσβλέπουν στην ευρωπαϊκή προοπτική και την ένταξη της Σερβίας. Από την δική μου πλευρά και σε ό,τι με αφορά είναι η τελευταία μου συμμετοχή και ευχαριστώ με την ευκαιρία τους Προέδρους και όλους εσάς. Μια σκέψη μόνο θα καταθέσω όσον αφορά την γενική συζήτηση και τις συζητήσεις που είχαμε στο παρελθόν. Στην Επιτροπή αυτή, ξέρετε, έχουμε κυρίως βουλευτές που υποστηρίζουν, υποστηρίζουν θερμά την μελλοντική ένταξη της Σερβίας. Όμως, πολλές φορές επιτελούμε άχαρο ρόλο. Ξέρετε, όταν συζητούμε και τις δυσκολίες, τα πιο κανθόδη, γιατί ερμηνεύεται η στάση μας ως επικριτική της Σερβίας. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ίσα ίσα θα υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κούκαν νωρίτερα, ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά, ας πούμε, στον τομέα της ελευθερίας του τύπου. Ε, είδατε τα αποτελέσματα της μελέτης της Freedom House. Αυτά δεν μπορεί να τα γνωρίσει κανείς. Ούτε μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι πρόκειται για άδικη μεταχείριση της Σερβίας. Αυτά μας λένε και οι πρεσβείες μας, αυτά μας λένε και άλλοι. Το ξέρουμε, ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Οπότε η παρατήρηση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή είναι. Είτε τη βλέπει κανείς άδικη, είτε όχι, αλλά κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν ε, αναφερόμαστε στην κατάσταση αυτή ως πρόσκομα, ως εμπόδιο. Όχι, πρόκειται για προαπαιτούμενο για την συνέχιση τη περαιτέρω πορεία. Αλλιώ λύση δεν θα βρούμε, αλλιώ δεν θα ανοίξουν περαιτέρω κεφάλαια. Δεν θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Γιατί αυτό είναι ο τελικό στόχο. Το πιο σημαντικό από όλα είναι οι αλλαγέ να ελοπιθούν στην πράξη, στην ελευθερία του τύπου, όσον αφορά την αντιπολίτευση, του θεσμού κλπ. Δεν θα συζητήσουμε εμεί εδώ. Ξέρετε, δεν μα πέφτει λόγο για, για την ιστορική πολιτική τη Σερβία, ε, για τι πολιτικέ αντιπαραθέσει. Η δημοκρατία όμω είναι αυτό. Είναι αντιπαράθεση, αλλά είναι και εξέβρεση συνένεση χάρη στου θεσμού που συναποτελούν την δημοκρατία. Κάθε φορά που διαφωνούμε. Οπότε το δικό μου μήνυμα είναι και δεν το απευθύνω ειδικά στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση. Το μήνυμά μου είναι απλό. Όλα αυτά τα θεσμικά προβλήματα πρέπει να επιληθούν με τρόπο που θα οδηγήσει στην επίτευξη συνένεσης. Από την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω να πω ότι και εμείς έχουμε εδώ κάθε είδου αντιπαραθέσεις και διαφορετικές ιδέες. Όμως, κανείς δεν αμφισβητεί το θεμητό, την νομιμότητα των θεσμών μας που δίνουν την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί. Κανείς δεν αμφισβητεί την νομιοποίηση των εκλογών. Πρόβλημα είναι μόνο όταν αρχίσουν να αμφισβητούνται οι δημοκρατικοί θεσμοί. Και γι' αυτό υπογραμμίζω αυτό που είπα. Ε, και το λέω ως ένας εξ αυτών που επαναλαμβάνω είναι υπέρ τη ένταξη της Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Κολομπιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Συμπρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι τη Αντιπροσωπεία, θα ήθελα να θίξω αρχικά το ζήτημα του διαλόγου μεταξύ Βελγαδίου και Πρίστινα από διαφορετική όμω οπτική γωνία. Θεωρώ ότι το να υποτάξουμε την διαδικασία ένταξη τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με την ρύθμιση των διαφορών μεταξύ τη Σερβίας και του Κοσμοπεδίου ε, είναι μείζον ασφάλμα από διάφορε απόψει. Πρέπει να επιθυμήσουμε ότι το Κοσμοπέδιο δεν αναγνωρίζεται ε, από πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ανεξάρτητη χώρα. Κύπρος, Ελλάδα, Σλοβακία και άλλοι. Το να λοιπόν αυτό το ζήτημα της ένταξης της Σερβίας από κάτω από την ε, διευθέτηση ζητημάτων ε, λοιπόν σε, με μια χώρα που δεν αναγνωρίζεται, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα πρέπει να επιληθεί το ζήτημα και μετά να αποτελέσει αίρεση για την ένταξη της Σερβίας, όχι το αντίθετο. Το κοσμοπέδιο και η μετόχια λοιπόν είναι ε, τμήμα της Σερβίας, ε, ιδίως και επειδή υπάρχουν και θρησκευτικοί δεσμοί πρέπει να υπενθυμίσω δυσάρεστα αλλά παρέτα πράγματα. Μόνο μετά την στρατιωτική επέμβαση πριν από 20 χρόνια που, έκανε, που δημιούργησε χιλιάδες θύματα, ε, τελικά ε, είδε το φως της ημέρας αυτή η ψευδοδημοκρατία του κοσμοπεδίου. Τότε είχε χαρακτηριστεί ε, τρομοκρατική οργάνωση, τώρα όμως βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα status quo. Είχαμε αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις και διάφορες ε, διακρίσεις, ακόμα και εκφοβισμούς με στόχο να ε, αποτρέψουν τους Σέρβους από το να ε, ασκήσουν τη θρησκευτική τους ελευθερία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά λοιπόν να γίνει ένας διάλογος μεταξύ Κοσμοπεδίου και Βελιγραδίου, όμως προεπαιτούμενο εδώ είναι μια βούληση και των δύο μερών που καλή την πίστη θα προσπαθήσουν να εξεύρουν λύσεις. Ε, αμοιβαία αποφελής και για τους δύο. Όμω αυτό δεν ισχύει σε αυτήν την περίπτωση και αυτό είναι προφανέ. Ο, ο Υπουργό θα υπενθύμησε προηγουμένω να πω και εγώ ότι πρόσφατα οι εντάσει μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα ε, εντάθηκαν ακόμα περισσότερο. Και έτσι η προπτική ενό επικοδηματικού διαλόγου απομακρύνεται, καθότι και στι 6 Νοεμβρίου το Κοσμοπέδιο ε, υιοθέτησε δασμούς 100% ε, κατά των ε, σερβικών ε, προϊόντων. Η κυβέρνηση του Κοσμοπεδίου φυσικά γύρισε την πλάτη στις κριτικές και επικρίσεις της διεθνούς κοινής γνώμης, ιδίως όταν στις 21 Νοεμβρίου η είπατε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Μογκερίνη, δήλωσε ότι η ε, επιβολή τέτοιων δασμών ε, αντιβαίνει στη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών ε, και στην Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοσμοπεδίου. Στη συνέχεια, σε ένα κλίμα αυξανόμενης έντασης, η Βουλή του Κοσμοπεδίου τον Δεκέμβριο υιοθέτησε ε, νόμο για την ασφάλεια του κοσμοπεδίου. Αυτός ο νέος νόμος ε, που διακήρυξε και ο πρόεδρος ε, προβλέπει την ίδρυση στρατού και αυτό θεωρώ ότι δικαίως θεωρείται απειλή από τη Σερβική Δημοκρατία και απειλή και προς την σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Όλα αυτά αποδεικνύουν την αδυναμία της ευρωπαϊκής διαπραγματικής ισχύω, δυστυχώς, και δεν υπάρχει καμία λύση που μπορεί να επιτευχθεί καλή τυπή σε αυτή τη στιγμή με το κοσμοπέδιο σε ό,τι αφορά και την προστασία των Σέρβων ε, του κοσμοπεδίου. Κλείνοντας, εγώ είμαι ειδικό απεσταλμένος ε, ε ο Σίντου Λαμινούκ ειδικό απεσταλμένο στο ΟΗΕ αναφέρει ότι στην Πρίστινα δεν υπάρχει ενιαία θέση για την κατάλληλη ε, θέση επανεκκίνηση του διαλόγου με το Βελιγράδι, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σημείο ρήξη τι τελευταίε ημέρε. Και υπάρχουν ε, μεγάλες ανησυχίες ότι αφορά την μελλοντική βιωσιμότητα του κυβερνητικού συνασπισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κοσμοπέδιο. Νομίζω ότι αυτή η αξιολόγηση πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερως, γιατί δεν, δεν αναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στη Σερβία για να ε, προστατεύσει την ακαιρεότητά της ε, ως έθνος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κολομιέ. Φτάνουμε στο τέλος ε, της συνεδρίασης. Θα επανέλθουμε στις 6. υπό τον αγαπητό συμπρόεδρο κύριο Όλιτς.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

samo u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

poštovani članovi zajedničkog parlamentarnog odbora nastavljamo sa radom pošto su diskusije nastavljene i po tačkom pod rednim brojem 3 i pod rednim brojem četiri nastavićemo ih na osnovu napravljene liste prijavljenih dajem reč gospodinu đuriću izvolite hvala poštovani kopredsedavajući gospodina Orliću i hvala i gospodinu Kukanu. Ja ću se truditi da maksimalno skratim ono što sam nameravao da kažem, obzirom da smo već dosta toga rekli i da je i agenda dosta, dosta Πολλά ακούσαμε προηγουμένω και είναι πληρέστατη μέρη στη διάταξη. Θα ήθελα λοιπόν να διαπιστώσω ότι στην κοινωνία μας ε, δεν υπάρχει δυστυχώς ε, ομοφωνία γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ συχνά ακούμε ότι τις μεταρρυθμίσει πρέπει να τι κάνουμε για λογαριασμό μας, ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχω να κάνω το εξή σχόλιο. Είναι σαν ένα φιλικό αγώνα στο ποδόσφαιρο, όπου τελικά δεν έχει και σημασία το αποτέλεσμα. Εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε οτιδήποτε είναι φιλοευρωπαϊκό, αλλά έχουμε ακόμα αρκετά, αρκετούς ευρωσκεπτικιστές, ακόμα και κάποιους που είναι ξεκάθαρα αντίθετοι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν και βήμα στα μέσα ενημέρωσης. Πολύ συχνά μάλιστα πρόκειται για μέσα ενημέρωσης που πρόσκυνται στην ε, κυβέρνηση, ακόμα και αν ε, οι ιδιοκτήτες τους ε, βρίσκονται στη Δύση. Υπάρχουν ε, φυσικά και άλλοι που είναι ιδιαίτερα θετικοί ως προς τη Ρωσία. Το οποίο φυσικά αποτελεί πρόβλημα και απειλή για τις φιλοδυτικές δυνάμεις. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την κατάσταση στο Κοινοβούλιο και τις διαδηλώσεις, καθώς και για την εκλογική διαδικασία. Η αντιπολίτευση μποϊκοτάρει αυτή τη στιγμή ε, το Κοινοβούλιο στη Σερβία και λένε μάλιστα ότι θέλουν να μποϊκοτάρουν και τις εκλογές. Ε, λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο κύριος Μακάλιστερ. Ακούσαμε όμως ε, τη δήλωση του για το Free Europe, όπου είπε ότι θα επανέλθει η αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο, γιατί εκεί πρέπει να οικοδομηθεί ο πολιτικός διάλογος. Συμφωνούμε απολύτως με αυτή τη θέση. Και μάλιστα κοινοποιήσαμε αυτή τη δήλωση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να λάβουν μεγαλύτερη προβολή. Λάβαμε πολλά σχόλια και είδαμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να περασπιστούμε αυτή τη θέση του κ. Μακάλιστερ, παρότι το προσπαθήσαμε. Το κλίμα όμως ε, στο Σερβικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή είναι και η αιτία του μποϊκοτάζ. Δεν είναι χωρίς εξήγηση λοιπόν αυτή η εξέλιξη. Θέλει λοιπόν να έρθει κανείς στο κοινοβούλιο για να δει ε, τι κλίμα επικρατεί. Γιατί υπάρχει ένα κλίμα εκφοβισμού στο κοινοβούλιο. Και μάλιστα ο πρόεδρος ε, του κοινοβουλίου συχνά το επικροτεί. Εμείς θέλουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Είμαστε το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης ε, που ε, συμμετέχει στις εργασίες του Κοινοβουλίου. Ήμασταν εκεί ε, στην έναρξη των ερηνών εργασιών και θέλουμε να τίνουμε μια χείρα συνεργασίας και βελτίωσης του κλίματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διαδηλώσεις, νομίζω ότι οδηγούν σε περαιτέρω πόλωση στη Σερβία, ενώ εμείς χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνένεση. Έχουμε την εντύπωση ότι οι δύο πλευρές δεν ε, καταβάλουν επαρκείς προσπάθειες για την εξομάλυνση της κατάστασης. Εμείς δεν θέλουμε και δεν είμαστε υπέρ της ε, βίαιης εισβολής ε, στη ραδιοτηλεόραση, όμως δεν μπορούμε να επιτρέψουμε και φαινόμενα όπως αυτά της, ε, των κομμάτων που είναι στην εξουσία που λένε ότι δεν θέλουν να συζητήσουν και να κάνουν διάλογο με την αντιπολίτευση. μπορεί ενδεχομένως να μην απαιτούμε κάτι τέτοιο από τον πρόεδρο ε, της Σερβικής Δημοκρατίας να διοργανώσει τέτοιο διάλογο. Ίσως ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου να πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι με την ε, ατμόσφαιρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην είναι πλέον δυνατό να διοργανώσουμε ένα τέτοιο διάλογο. Γιατί ορισμένοι σήμερα θεωρούν ότι δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το διάλογο στο Κοινοβούλιο μεταξύ της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Το εκλογικό σύστημα παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν υπάρχει κάποια παρατυπία που θα μπορούσε να επηρεάσει ε, το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά υπάρχουν πολλές παρατυπίες πριν από τις εκλογές. Η Transparency International και άλλε μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, έχουν επισημάνει τα κακό κείμενα. Και σε ό,τι αφορά την προεκλογική εκστρατεία, έχουμε εκπροσώπους της κυβέρνησης που προβάλλουν ε, το πολιτικό τους ε, κόμμα. Άλλοι έχουν προσληφθεί στο δημόσιο επειδή ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο κόμμα. άλλοι χρησιμοποιούν ε, δημόσιους εξωματούχους για να προβάλλουν ε, την προεκλογική τους εκστρατεία. Υπάρχουν άλλοι που εκφοβίζουν ε, το εκλογικό σώμα. Και σε επίπεδο νομικού πλαισίου υπάρχουν αδυναμίες και θα πρέπει να επανεξεταστεί. Απειλείται ο δημόσιος διάλογος. Οι πολίτες λοιπόν στη Σερβία δεν γνωρίζουν αυτά που συζητούμε εδώ σήμερα. Ακούνε μόνο τι κάνει ο πρόεδρος, αν επισκέφθηκε το τάδε χωριό, αλλά κατά τα λοιπά δεν γνωρίζουν τίποτα. Όταν επελέγει ο διαμεσολαβητής στη Σερβία, ε, δεν ενημερώθηκε η κοινή γνώμη για το τι, ποια είναι τα καθήκοντα, ε, πώς μπορούν ε, να αποταθούν σε αυτό το πρόσωπο, δεν ε, έμαθαν τίποτα. Και άλλα προβλήματα υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς και τα καθήκοντά τους, που επίσης δεν είναι σαφώς προσδιορισμένα, τους δικαστικούς κλητήρες μάλλον, είναι πραγματικό πρόβλημα στη σερβική κοινωνία γιατί υπάρχουν και πολλά αυθαίρετα κτίσματα. Πολλά μένουν ακόμα να γίνουν λοιπόν εκεί. Και τέλος έχουμε και το οικονομικό πρόβλημα του brain drain. Πολλοί κόσμος που φεύγει λοιπόν από τη Σερβία. Το καλύτερο, τα καλύτερα μυαλά τη σερβία ε, έχουν ήδη ε, πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορώ να πω σε όσου φοβούνται την ένταξη τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να εξετάσουμε και τη διακήρυξη. Εγώ λοιπόν να σας πω ότι δεν θα πάρω το λόγο, αλλά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα μιλήσω για τη σχέση μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Θεωρώ ότι υπάρχει η εξή λύση. Να επιλύσουμε τα κοινωνικά και άλλα προβλήματα που έχουμε σε αυτές τις περιοχές. Αυτό ισχύει για όλους. Ποιο είναι το μείζον πρόβλημα και στο Κοσμοπέδιο Μετόχια και στη Σερβία. Ε, ψωμί, ειρήνη, και εργασία. Αυτά τα τρία προβλήματα πρέπει να επιληθούν και θα μας επιτρέψουν να ξεχάσουμε τα υπόλοιπα ή τουλάχιστον να τα θέσουμε κατά μέρος. Γι' αυτό και πρέπει να εργαστούμε για τη γνώση, για τη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση των εγωιστικών τάσεων. Στην κοινωνία μας έχουμε τους πολύ πλούσιους που ζουν πλουσιοπάροχα, ενώ η πλειονότητα του κόσμου ζει με τα πολύ λίγα. Πρέπει λοιπόν να εξομαλύνουμε αυτές τις διαφορές και να εκπαιδεύσουμε αυτούς που έχουν πάρα πολλά, ούτως ώστε να βοηθήσουν τους ε, πιο αδύναμους. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έδινε, επένδυε σημαντικά ποσά στη Σερβία, θα ξεχνούσαμε όλα μας τα προβλήματα. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά το κοσμοπαίδιο, ουσιαστικά κάνει τα στραβά μάτια. Κάνει ότι δεν βλέπει το πραγματικό πρόβλημα. Η συζήτηση με τον κύριο Κολομπιέ μου έδειξε ότι υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν διαφορετικά το πρόβλημα. Και ελπίζω στο μέλλον όλοι μαζί να έχουμε το θάρρος να επιλύσουμε με πολιτισμένο τρόπο αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ κύριος Μιγιάτοβιτς. Εγώ θα είμαι ακόμη πιο σύντομος όπως Λιμπισσά, Τα περισσότερα ελέγχθησαν όσον αφορά τον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινες. Σύμφωνα με τα περισσότερα δεν θα τα επαναλάβω. Όμως είναι σημαντικό το ότι σήμερα έχει παγώσει ο διάλογος. Δεν υπάρχει διάλογος. Πώς θα τον ε, επαναδρομολογήσουμε. Το είπαμε. Προϋπόθεση είναι η εξάλληψη των δασμών 100% για τα εμπορεύματα από Σερβία. Μετά συνεχίζουμε. Διότι στη Σερβία ε, δεν αρέσει αυτή η τελμάτωση. Και θα θυμίσω αυτό που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να είμαστε όμοιρος του κοσμοπεδίου. Το που ο συνάδελφος τέλει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυναμεί. Προσπαθεί, έχει καλή θέληση, όμως η Πρίστινα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ακριβώς για να μην εξευρεθεί λύση αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω. Ίσως χρειάζεται περισσότερη πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πρίστινα και ενδεχομένως να διαχωριστεί η δική μας ένταξη από τον διάλογο με την Πρίστινα. Γιατί ο διάλογος θέλει δύο. Τώρα η περαιτέρω όξυνση της κατάστασης και στο, στα βόρεια και στα νότια του Κωσόβου όπου έχουμε σερβικούς πληθυσμούς οι οποίοι ζουν υπό το κράτος του φόβου. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια παγιωμένη κατάσταση που θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε να έχουμε λόγο στην επίλυση του προβλήματος. Θα ήθελα επίσης να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τον κύριο Κούκαν. Γίναμε φίλοι με τον καιρό. κ. Κούκαν, όχι εδώ σε αυτήν την επιτροπή, αλλά σε άλλους χώρους έδειξε ρεαλισμό και υποστήριξε την υποψηφιότητά μας. Σας ευχαριστώ κύριε Κούκαν και προσωπικώς γιατί νομίζω πετύχαμε πολλά μαζί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5 συστάσεις. Έχουμε έναν πίνακα εν προκειμένου με τα σχόλια των δύο συμπροέδρων. Είναι πράγματα που συζητήσαμε και με τις δύο αντιπροσωπείες κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Αυτή τη στιγμή το κείμενο μεταφράζεται στα σερβικά. ειδοποιώ τους διερμηνείς ότι θα διαβάσω και στα σερβικά και στα αγγλικά. Οπότε, διερμηνία υπάρχει, νομίζω θα τα καταφέρουμε για να δείτε τι ακριβώς προκρίναμε. Ας παρακολουθεί και η γραμματεία. Πείτε μου αν υπάρχει κάποιο λάθος, παρακαλώ. Έχουμε κάποιες τροπολογίες. Εγώ, Ντέλη, Ορσίτς, Στεμίροβιτς, Χόβατς, Ορλίτς. Έχουμε εδώ μερικές τροπολογίες όπως έλεγα. Όπως βλέπετε, έχουμε νέες διατυπώσεις αποτέλεσμα του συμβεσμού των δύο αντιπροσωπιών και άλλων. Παράγραφος 1, δύο τροπολογίες. Μαρινά Άντερσον. Εδώ δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε. Μιγιάτοβιτς συμφωνούμε. Εκεί βρήκαμε συμβαστική λύση, βλέπετε το περιεχόμενο. Ω μια προτεραιότητα και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την δέσμευσή τη προ την κατεύθυνση αυτή, λέει το κείμενο. Οπότε και εδώ συμφωνούμε. Οι δύο αντιπροσωπείε. Υπάρχει κανένα σχόλιο. Πολύ ωραία. Έγκρινεται η τροπολογία. Παράγραφος 2. Δύο τροπολογίες. Γραπτές και οι δύο. Είναι τρία και τέσσερα, Φλέκενστάιν, Πίτσουλα, Άντερσον, αυτή γίνεται δεκτή. Και η τέσσερα, Μαριανοβίτς, Άντερσον και αυτή δεκτή. Παρακαλώ κάποιο σχόλιο. Όχι. Πολύ ωραία και οι δύο τροπολογίες εγκρίνονται. Παράγραφος 3. Δύο τροπολογίες και αυτές υποβλήθηκαν γραπτός, οι 5 και 6 από την Σερβική Βουλή. Με καμία δεν συμφωνήσαμε. Έχουμε όμως μία προφορική τεχνικής φύσεως. Αποτελεί διόρθωση στο κείμενο. Την διαβάζω. Εκεί που λέει και συνεχίζει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Τα μέτρα αυτά, τα οποία παραβιάζουν το πνεύμα της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Και μετά το κείμενο συνεχίζει χωρίς περαιτέρω αλλαγή. Νομίζω ότι εδώ καταφέραμε να συμφωνήσουμε. Συμφωνούν και οι δύο συμπρόεδροι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σχόλια ε, για την παράγραφο 3. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Η προφορική λοιπόν τροπολογία που μόλις διάβασα αποτελεί πλέον ε, μέρος του κειμένου. Υπέρ και 6 απορρίφθηκαν. Παράγραφος 4, τροπολογία 7 και τροπολογία 8. Και εδώ δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει επισχόλιο. Όχι. Οπότε οι τροπολογίες αυτές απορρίπτονται. Παράγραφος 5, τροπολογίες 9, 10, 11 και 12. Και εδώ δεν συμφωνήσαμε. Ε, με καμία από αυτές, δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να μιλήσει. Όχι. Οπότε, επαναλαμβάνω, οι τροπολογίες αυτές απορρίπτονται. Παράγραφος 4 μία τροπολογία στην 6 με συγχωρείτε και θα απορρίπτεται παράγραφος 7 τροπολογίες 14 και 15 ούτε δεν υπάρχει συμφωνία θέλει κανείς το λόγο όχι οι τροπολογίες λοιπόν αυτές απορρίπτονται για τη νέα παράγραφο 7α, την οποία προτείνει ο κ. Βλέπετε το κείμενο εδώ, στα αγγλικά. Εδώ πρόκειται περί σύμπηξη αυτή με την 25, στην προτελευταία σελίδα. Προτείνουν Νικόβατ και Όρλιτς. Πρόκειται νέο κείμενο λοιπόν που θα αποτελέσει αν, γίνει, αν εγκριθεί την παράγραφο 7α. Είναι κοινό κείμενο. Οι δύο συμπρόεδροι συμφώνησαν, συμφωνούμε όλοι πολύ ωραία. Οπότε προστίθεται νέα παράγραφος 7α. Η γραμματεία θα επαναρρυθμίσει τα, τις παραγράφους. Παράγραφος 8 Παράγραφος 17 και 18 λέει ο μιλητής. Καμία δεν συνομολογήθηκε από τους συμπροέδρους. Έχουμε και μία προφορική όμως. Στην παράγραφο 8. Σύμφωνα με αυτή πρέπει να αφαιρεθούν τα εισαγωγικά. Μα ξέρετε πρόκειται για παράθεμα, γι' αυτό υπάρχουν εισαγωγικά. Η πρόταση είναι να αφαιρεθούν τα εισαγωγικά. Συμφώνησαν οι δύο αντιπροσωπείε, συμφωνήσαμε όλοι, πολύ ωραία. Η προφορική λοιπόν αυτή περιφέρεση των εισαγωγικών γίνεται δεκτή. Οι γραπτές τροπολογίες, όπως προείπα, απορρίπτονται. Παράγραφος 9. Εδώ είναι 18. Και στη 10 έχουμε τις 19 και 20. Συμφωνούνται και, και οι δύο. Γίνονται αποδεκτέ και οι δύο. Θέλει κανεί να μιλήσει, όχι. Α, με συγχωρείτε, η 19 λέει ο μιλητή απορρίπτεται. Παράγραφος 11, τροπολογία 21. Προτάθηκε από τον κύριο Χακμαρ. Οι συμπρόεδροι προτείνουν να γίνει υποδεκτή. Με ένα συμβεστικό κείμενο, το οποίο αφορά τροποποίηση της τροπολογίας. Έχουμε λοιπόν μια συμβαστική, η οποία έχει ως εξής όσον αφορά τις υφιστάμενες εισαγωγές αερίου. Με αυτή τη διόρθωση. Η τροπολογία λοιπόν του κυρίου Χέκμαρκ γίνεται αποδεκτή. Εγκρίνεται με αυτήν την μικρή τροποποίηση, παρακαλώ. Α, αυτό είναι το κείμενο ε, και δεν λέει πλέον στο ρωσικό, στις ρωσικές εισαγωγές αέριο. Ωραία, κατάλαβα. Θέλει κανείς άλλος να μιλήσει. Η τροπολογία αυτή λοιπόν, με τη μικρή αυτή αλλαγή, γίνεται αποδεκτή. Παράγραφος 12, τροπολογία 22. Και εδώ έχουμε διαφωνία των συμπρόεδρων απορρίπτεται. Παράγραφος 13, τροπολογία 23. Ούτε δεν υπάρχει συμφωνία. Κάτι θέλει να μιλήσει. Απορρίπτεται. Παράγραφος 15, τροπολογία 24. το κύριο Στοημίροβιτς, οι συμπρόεδροι συμφωνούν. Θέλει κανείς να μιλήσει. Πολύ ωραία, εγκρίνεται. Η 24 λοιπόν εγκρίνεται. 25 τώρα. Εγκρίθηκε όπως εξήγησε προηγουμένως. Ενσωματώνεται στο νέο κείμενο της 7α μαζί με αυτό το οποίο πρότεινε ο κ. Τέλη. Άρα κλείσαμε και με αυτό. Και πάμε στην τροπολογία 26 της κ. Κόβατς. Συμφωνούν οι συμπρόεδροι με μία μικρή διόρθωση. Τη διόρθωση τη βλέπετε στο έγγραφο μπροστά σας. Τονίζει, διαγράφουμε το Regatta Principle και με άλλες δύο μικροδιορθώσεις η τροπολογία αυτή γίνεται δεκτή. Οπότε, θέλει κανείς το λόγο. Η τροπολογία αυτή είναι και αυτή μέρος του ανακοινοθέντος με τη μορφή νέας παραγράφου, όπως είπα. Η γραμματεία θα αριθμίσει εκ νέου το κείμενο, τις παραγράφους του κειμένου. Παρακαλούθησα πολύ προσεκτικά, αν και δεν ήταν εύκολο. Θέλω να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Α, ο κ. Τελή με ακούει και νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου, τον βλέπω να χαμογελάει. Κύριε Συμπρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και μια τελική ψηφοφορία. Το ερώτημα θα είναι ποιος είναι υπέρ, ε, ποιο είναι υπέρ ε, του τελικού κειμένου, όπως τρόπο θα ενισχύει. Εγώ ψηφίζω ναι. Ευχαριστώ κύριε Κουκάν. Ε, Σύμφωνα με εσάς. και ευχαριστώ που μεταφέρετε και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε, ποιο είναι ε, υπέρ του κειμένου από το Σερβικό Κοινοβούλιο. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Πολύ ωραία. Οπότε συνάγω ότι και οι δύο αντιπροσωπείες ε, εγκρίνουν το τρόπο είναι κείμενο. Στα διάφορα τώρα, που είναι και το τελευταίο σημείο της μίλησης διάταξης, θέλει κανείς να μιλήσει στο πλαίσιο του σημείου 7. Α, επόμενη συνεδρίαση. Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, 30-31 Οκτωβρίου, στο Βελιγράδι. Θέλει κανείς από την άλλη ημερομηνία. Όχι. Από ό,τι βλέπω. Οπότε, ευχαριστώ όλες και όλους. Α, ο λόγος του κ. Κούκαν κύριος ε, Ντέλη μας έφερε. Είδα ότι πήρε καφέ, οπότε να συνεχίσουμε τη συζήτηση για να μπορέσει να τον απολαύσει. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μας εργασιών. Χαίρομαι που καταφέραμε να υιοθετήσουμε την ε, κοινή διακήρυξη. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό κείμενο. Και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Εκτιμώ ιδιαίτερως ε, τα καλά σας λόγια και πάντα είναι ευχάριστο να ακούει κανείς ε, επένους, αλλά εγώ το ερμηνεύω ως μια υποχρέωση να συνεχίσω να εργαζόμαι για τη Σερβία και για εσάς. Ήμουν ε, στο γραφείο μου προηγουμένως και κοιτούσα τις ε, φωτογραφίες. Είμαστε όλοι νέοι, αλλά ξέρετε το χρόνο δεν το σταματάει κανείς. Έχουμε όλοι ωραίες αναμνήσεις και θα έχουμε ωραίες αναμνήσεις. Ευχαριστώ. Το δώρο αυτό είναι πολύ ωραίο. Ξέρετε, όλα αυτά θα μας θυμίζουν ωραία πράγματα θα μας θυμίζουν ε, ωραίες στιγμές και είχαμε πολλές ωραίες ε, στιγμές. Φάμε τις ε, συζητήσεις. Ήταν ωραία ακόμα και όταν διαφωνούσαμε, αλλά αυτό είναι φυσικό. Ξέραμε πάντως σε κάθε περίπτωση ότι είχαμε ένα κοινό στόχο. Και είναι κοινό μα καθήκον να βοηθήσουμε τη Σερβία στην ευρωπαϊκή της προοπτική στο μέλλον. Σας ευχόμαστε λοιπόν ε, ό,τι καλύτερο. Θα έρθω στο Βελιγράδι και θα σας επισκεφθώ. Παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη να πιούμε ένα καφέ όταν έρθω. Γιατί ασχολούμαι με τα Δυτικά Βαλκάνια εδώ και πολλά χρόνια. Ε, και με κάθε μετριοπάθεια μπορώ να σας πω ότι ξέρω λίγα πράγματα πλέον για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και μια τέτοια γνώση δεν γίνεται να την πετάξουμε στο κάλαθο των αχρήστων, πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να την καλλιεργήσουμε λοιπόν και ελπίζω να με βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιστροφή, συνεχίστε το έργο σας, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους τους τομείς. Καλή τύχη και στο επανειδήν.